Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε δέκα ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλούς ευρωβουλευτές που είναι έξω στο διάδρομο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να αρχίσουμε και να ψηφίσουμε. Η συγγήτρια είναι η κυρία Πατρίτσια Τόγια. Ας αρχίσουμε. Σχέδιο έκθεσης για την ε, πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων 700 MHz στην Ένωση. Συνεπώς, πρόκειται για το φάσμα. Αρχίζουμε λοιπόν με μια δοκιμή στην ψηφοφορία, όπως κάνουμε πάντα. Ψηφίστε παρακαλώ. Εντάξει. Το αποτέλεσμα μερικό σα ικανοποιεί στι ΗΠΑ, ρωτάει ο πρόεδρο. Ψηφίστε όμω τώρα. Πέρα τη ψηφοφορία αυτή τη δοκιμαστική. 21%. Δεν ξέρω, 12 είναι μερικώς ικανοποιημένοι καθόλου, δύσκολα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 Έτσι είχα ενημερωθεί ότι είχε αποσυρθεί. Εγώ φταίω που δεν σας ενημερώσα από αυτού. Οπότε σεβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σεβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σεβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σεβαστική 8, 1, αναφορική σκέψη 1, κατά Α, ναι, ξέχασα. 203, τροπολογία 203 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα σεβαστική 8, αιτιολογική σκέψη 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σεβαστική 9, αιτιολογική σκέψη 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10, αιτιολογική σκέψη 2α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11, αιτιολογική σκέψη 2β υπέρ,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 Αιτιολογική σκέψη 16 τώρα. Τροπολογία 132-133 μαζί για την ίδια Σιπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, ας ελέγξουμε. Να ελέγχουμε που και που ηλεκτρονικά. 134 λοιπόν. Μπορείτε να ψηφίσετε. Α, όχι. Μια στιγμή. Ψηφίζει ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω ψηφίζει. Τώρα εντάξει. Ωραία, τώρα πέρα τη ψηφοφορία και το αποτέλεσμα σαφώς απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία Ονομαστική ψηφοφορία βέβαια. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πάλι ένας από το ΕΛΚ παραπάνω ψηφίζει. Τώρα είναι εντάξει. Πέρα της ψηφοφορίας. Σαφώς εγκρίνεται η έκθεση αυτή. Τώρα νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα, πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε τις ε, διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ωραία. Εγκρίνεται επίσης Κυρία Τόγε, η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα λεπτό θέλω για να ευχαριστήσω όχι επίσημα και τυπικά αλλά από καρδία σε όλους εκείνους που εργάστηκαν αυτό το αποτέλεσμα πιστεύω το οποίο είναι ισορροπημένο αποτέλεσμα και αυτό είναι το καλύτερο, ένα αποτέλεσμα ισορροπημένο. Ευχαριστώ τους Κιώδης, ξεκινώντας τον συνάνθρωπο Όκμαρ, όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής όμως οι οποίοι προσπάθησαν να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και το προσωπικό μας, του γραφείου μας και όλων των σκιωδών που συνεργάστηκαν. Ευχαριστώ. Thank you, Σας ευχαριστούμε. πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Και την εισηγήτρια και όλους τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέρφους. Ωραία, τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Σημείο 13. Πρόκειται για το ελεγκτικό συνέδριο και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Άλεξ Μπρένικ που είναι μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε? Mm. Σας παρακαλώ. Καθίστε, κύριε Μπρένικ Μάιερ, καλώς ήρθατε. Το το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την ετήσια έκθεσή του για το 2015. Αυτό είναι το θέμα μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ. Σταματήστε τις συζητήσεις εδώ μέσα και τα πηγαδάκια. Αλλιώς, αν θέλετε να συνεχίσετε τα πηγαδάκια, εκτός αιθούσης. Ή σταματάτε τώρα μέσω τη συζήτηση ή Λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Μπρένικ Μάιερ είναι υπεύθυνο για το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στο λεκτικό συνέδριο. Το 2014 έγινε μέλος του λεκτικού συνεδρίου. Ήταν ε, ο συνήγορος του πολίτη στην Ολλανδία πριν και ε, υπεύθυνο σε διάφορα δικαστήρια, όπως για παράδειγμα το διοικητικό στην Ολλανδία. Πολύ σημαντική θέση. Έχει και μακρά ακαδημαϊκή σταδιοδρομία έχει δοκτορά φιλοσοφίας από το Τίλμπουργκ και είναι επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Για μας που είμαστε στην Επιτροπή Ήτρε, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι πιστεύει το ελεγκτικό συνέδριο για τα κεφάλαια της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, για, τον, για το Horizon 2020 για παράδειγμα. Ο κύριος Μπρένικμαγερ, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω τι γίνεται με το κεφάλαιο 5 στην ετήσια έκθεσή μας όσον αφορά τα θέματα που σας απασχολούν. Θα είμαι σύντομος και θα υπογραμμίσω ένα σημαντικό θέμα. Και αυτό είναι η καινοτομία στους ελέγχους. Στην εισαγωγή μου λοιπόν θα ξεκαθαρίσω γιατί η καινοτομία στον έλεγχο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως όσον αφορά το Horizon 2020. Ξέρετε ότι η καινοτομία είναι μέρος βέβαια του προγράμματος αυτού, ορίζοντας 2020. Θα αρχίσω λοιπόν με τα κύρια θέματα με τα οποία θα ασχοληθώ. Γιατί δεν συμμορφώνονται οι δικαιούχοι και σε τι θα βοηθήσει η καινοτομία αυτή. Το δεύτερο μου θέμα είναι γιατί δεν συμμορφώνονται οι δικαιούχοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω. Συνεπώς, τι βλέπουμε. Το πλαίσιο για τον ορίζοντα 2020 έτσι καλώς αποτελεί βελτίωση του προγράμματος πλαισίου 7. Και η έκθεσή μας καλύπτει σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα ακριβώς αυτό πλαίσιο 7. Αυτό εξετάζουμε λοιπόν. Και την επόμενη χρονιά και την μεθεπόμενη θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για ε, το νορίζοντα 2020. όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για τη μη συμμόρφωση, το ποσοστό σφάλματος είναι 4,4% το 2015. Το 2014 ήταν 5,6% και το 2013 ήταν 4%. Το ερώτημα είναι, πρόκειται για βελτίωση ή όχι. Και εγώ έχω ανάμεκτα συναισθήματα για να σας απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Γιατί καταρχήν μπορούμε να πούμε, ζήτω η Ευρωπαϊκή πέτυχε και μείωσε το ποσοστό σφάλματος από το 5,6 στο 4,4. Αλλά από την άλλη, έχω την αίσθηση ότι η αλλαγή αυτή δεν είναι σημαντική. Συνεπώς του χρόνου μπορεί να είναι 6% το σφάλμα. Και αν τότε με ρωτήσετε, είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό για την Επιτροπή, θα σας πω όχι, γιατί τελικά τα ποσοστά αυτά σύμφωνα με τη μεθοδολογία μας, οι αλλαγές δηλαδή, δεν είναι τόσο ουσιαστικές. Οπότε ερχόμαστε σε ερώτημα πώς να καινοτομήσουμε το έργο του ελεκτικού συνεδρίου αφενός και της ελεκτικής ομάδας της Κομισιόν από την άλλη, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ρώτησα λοιπόν τους ελεκτές μας και η απάντηση στην ερώτηση του τι συμβαίνει στον τομέα αυτό της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνιστικότητας κτλ. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δέκα συναλλαγές για το κεφάλαιο 5 συνεισφέρουν σε 77% του συνολικού εκτίμησης σφάλματος. Αυτό σημαίνει ότι για το 4,4% 3,8% οφείλεται σε 10 μόνο περιπτώσεις το σφάλμα αυτό και μπορώ να σας τις απαριθμίσω τις περιπτώσεις αυτές. Θα βρείτε δύο όπου εμείς υποψιαζόμαστε ότι κάτι πραγματικά στραβό υπάρχει και ήρθαμε σε επαφή με την Όλαφ για αυτά, αλλά τα κύρια ζητήματα, τα υπόλοιπα, έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις δαπανών. Και ακριβώς Εκεί είναι το κόστος, για παράδειγμα, του προσωπικού που περιλαμβάνεται στα προγράμματα. Και άλλο σφάλμα, πολύ συχνό, είναι ότι νοικιάζονται εξωτερικοί consultants για τέτοια προγράμματα. Αυτοί οι σύμβουλοι, λοιπόν, θεωρούνται εσωτερικοί ή εξωτερικοί. Οπότε, έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα που είναι κατά των κανόνων, γιατί δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε εδώ πέρα το κόστος εξωτερικών συμβούλων. Αν λοιπόν θέσουμε το ερώτημα γιατί υπάρχουν σφάλματα, εντοπίζουμε για το 75% αυτό, το 77% αυτό που σας είπα, μπορούμε να έχουμε πέντε κατηγορίες αιτιών. Και έρχομαι στο επόμενο δεν βλέπουμε το δάσος και βλέπουμε το δέντρο. Δηλαδή ελέγχουμε τους κανόνες, προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι με τους κανόνες και τον έλεγχό τους και μετά προκύπτει ένα ζήτημα, ένα ε, μοντέλο συμφωνίας για παράδειγμα για το 2020. Αν μιλήσω με ερευνητέ, τι λένε, ένα μοντέλο συμφωνίες 700 σελίδες περίπου. Το υποβάλλουμε, το μαθαίνουμε. Έχουμε βέβαια διάφορα περίπλοκα διεθνή προγράμματα, 700 σελίδες, έτσι. Και το πρόβλημα είναι η δυσπιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει. Γιατί αν αποκλείσετε από τους κανόνες, τότε είσαστε ύποπτος για απάτη. Και αυτό με φέρνει και στην επόμενη παρατήρησή μου. Το γιατί. Γιατί οι δικαιούχοι δεν συμμορφώνονται. Αυτή είναι μια συζήτηση που την είχα και με την Επίτροπη και με την Επίτροπο Γεώργιεβα και με το προσωπικό της Επιτροπής και με δικαιούχους του Horizon 2020 και του προγράμματος πλαίσιο 7. Γιατί λοιπόν οι δικαιούχοι δεν συμμορφώνονται. Δύο είναι οι απαντήσεις εδώ. Κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Είναι ένα μικρό ποσοστό, δεν θέλουν. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Κάνουν σφάλματα, όχι όμως από πρόθεση. Συνεπώς, σε αυτό τον τομέα, και εδώ είναι που έρχεται η καινοτομία, η καινοτομία είναι αναγκαία. Η καινοτομία στον έλεγχο. Είναι μια πολύ σημαντική προσέγγιση. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με πολύ κόσμο και λέμε είμαστε επαγγελματίες. Δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα σφάλμα. Συνεπώς θέλουμε και πρέπει να έχουμε νομική βεβαιότητα. Αν δηλαδή απαντήσω σε ένα πρόγραμμα η δήλωση δαπανών πρέπει να είναι σωστή και να γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος για το έργο μου. Έτσι σκέφτεται ο δικαιούχος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι δικαιούχοι να μάθουν από τα σφάλματα και η Επιτροπή να μάθει από τα σφάλματα και τα προγράμματα αυτά, το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και το Horizon 2020, να συνεχιστούν. Το σύστημα, μάλλον, εκταμίευσης κινδυνεύει να οδηγήσει σε σφάλματα όπου συμπληρώνεται, βάζει τα προσωπικά, το προσωπικό κόστος κτλ. Όλα αυτά κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε σφάλματα και τα, η προσέγγιση κατά αποκοπή μπορεί να βοηθήσει περισσότερο ή ένα σύστημα δικαιωμάτων. Αλλά αυτό μας φέρνει στο ότι μπορούμε με τον ορίζοντα 2020 να συνδέσουμε δικαιώματα για να διευκολύνουμε το σύστημα εκταμιεύσεων. Η νομική βεβαιότητα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχουμε πολλά στρώματα ελέγχων. Αρχίζουν στο επίπεδο πανεπιστημίων ή ομάδας πανεπιστημίων που έχουν ε, τους δικούς τους ελεκτές. Η ομάδα επίσης, το Ελεκτικό Συνέδριο επίσης έχει τους δικούς του ελεκτές και όλοι αυτοί από την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, τρίτη κτλ. κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν και εφαρμόσουν τους κανόνες με τον ίδιο τρόπο. Συζητάνε και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προδεύσει πολύ εισάγοντας το κέντρο στήριξης για να στηρίζει τους δικαιούχους στις δηλώσεις τους και στην ερμηνεία των κανόνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για παράδειγμα, ένα παράδειγμα από τη Γαλλία έχει να κάνει με την επιλεξιμότητα των προσωπικών δαπανών. Απ' τη μια είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στους κανόνες. Από την άλλη μεριά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες διαφωνίες υπάρχουν. Πού πρέπει να πάω, δεξιά, αριστερά, κάτω, στο έντυπο. Και οι συνέπειες απορρέουν από την πολυπλοκότητα του κανόνα. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, τη νομική βεβαιότητα και το, έμεσο κόστος. Στον ορίζοντα 2020 υπάρχει βελτίωση με την έννοια ότι οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 25% έμεσο κόστος κατά αποκοπή και βασίζονται σε δηλώσεις. Και τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει τάση στο σύστημα, μπορείτε τη χρηματοδότησή σας να την μεγιστοποιήσετε, και να πάρετε όσο γίνεται περισσότερα για το άμεσο κόστος και να ελαχιστοποιήσετε το υπόλοιπο. Οπότε μερικές φορές μπερδεύετε το ένα με το άλλο και τελικά στον ηλεκτρισμό, οι λογαριασμοί ηλεκτρισμού. Εκεί μπερδεύεται το άμεσο με το έμεσο κόστος ενώ χρειάζεστε διαφορετική απόδειξη για το ένα κομμάτι ηλεκτρισμού που ξοδέψατε και για το άλλο. Αλλά γι' αυτό ακριβώς εδώ υπάρχουν παρεξηγήσεις και οδηγούμαστε σε σφάλματα. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα μόνο του τι μπορεί να προκύψει. Και έρχομαι εδώ στο τέλος, δηλαδή τι ευκαιρίες υπάρχουν για τη βελτίωση του συστήματος. Υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά ζητήματα. Η αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών, η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλησίου και η ενδιάμεση αναθεώρηση του ορίζοντα 2020. Και έτσι έρχομαι στο επόμενο. Και αυτή ήταν και η δυσκολία μου με τον Επίτροπο Μαντέας. Μουέντας και την κυρία Γιώργεβα. Λοιπόν, ποιο είναι ο στόχο, ποια είναι η βάση μάλλον του ελέγχου. Η βάση του ελέγχου είναι κοινή λογική κυρίε και κύριοι. Γιατί αν ρωτήσετε έναν ελεγκτή ποια είναι η βάση αυτού που κάνει, θα σα πει είναι κοινή λογική. Και οι ελεγκτές την κοινή αυτή λογική τη βάζουν στου κανόνε. Και το επόμενο βήμα είναι ότι εφαρμόζουμε αυτού του κανόνε. Και εφαρμόζουμε αυτού του κανόνε πολύ αυστηρά. Και πολύ καλά κάνουμε και πολύ καλά γίνεται αυτό και μπορείτε να ελέγξετε έτσι αποτελεσματικά τις δαπάνες. Στο τέλος όμως, πάντα παραμένει το ερώτημα, τελικά αυτό που έχουμε κάνει είναι κοινή λογική. Και εγώ το ρώτησα και τον κύριο Μέντας και την κυρία Γιώργεβα, αν ελέγχουμε κάποιους τομείς πολιτικής τελικά εφαρμόζουμε την κοινή λογική. Γιατί αυτό είναι το κύριο ζήτημα που απασχολεί και τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουν νόημα όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή, και ήδη το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να κοιτάξουμε τις επιδόσεις. Πέρα από τη συμμόρφωση, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να δούμε τις επιδόσεις. Για να εφαρμόσουμε την κοινή λογική. Οπότε η έκκλησή μου είναι στους δημοσιονομικούς κανονισμούς, σας παρακαλώ, βάλτε ένα άρθρο 0 που να λέει ότι πάντα πρέπει να εφαρμόζεται κοινή λογική. Και η Κομισιόν τι λέει, η κοινή λογική τελικά δεν είναι και τόσο κοινή, ξέρετε. Η ανανομικό ζήτημα προκύπτει. Πώς εφαρμόζεται η κοινή λογική, με τι κριτήρια. Και έχω την αίσθηση ότι τελικά μερικοί δεν καταλαβαίνουν τι είναι η κοινή λογική. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί δεν πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, αλλά υπάρχουν βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μερικά τεχνικά στοιχεία, η ετήσια έκθεση του 2015 του Ελεκτικού Συνεδρίου δημοσιεύτηκε πριν από ένα μήνα και αναφερόμενοι στο πώς εφαρμόζεται ο προϋπολογισμός ανέφερε ότι υπάρχουν σφάλματα στις πληρωμές υπάρχει πρόβλημα αποτελεσματικότητα σε διάφορα συστήματα και το πιο ουσιαστικό για την επίτευξη αποτελεσμάτων όπως ορθά είπατε βγάζει νόημα, εξέρχεται νόημα. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η έκθεσή σας για το πρόγραμμα πλαίσιο 2020 που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και επίσης στο, στο κεφάλαιο 5 η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχολήσεως. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και εμάς όπως είναι Horizon 20, το Connecting Europe Facilities κτλ. Όλα αυτά είναι κεφάλαια τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα να συζητήσουμε μαζί σα το θέμα αυτό. Ο κύριος Έλεα από την ομάδα του ΕΛΚ. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όχι μονάχα διότι αυτό είναι η φόρμουλα αυροφροσύνης η οποία χρειάζεται, αλλά γιατί εσείς έχετε ανοίξει και ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επειδή το αναφέρατε, <clears throat> θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά που έκανε το Ελεκτικό Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας που βρισκόμαστε τώρα στη φάση της ε, εφαρμογής της ε, ε, αρχής λειτουργίας αυτού του Ινστιτούτου που θα μπορούσε πράγματι να ξεκινήσει πραγματικά να υπάρξει μια τομή σε αυτήν την λειτουργία αλλά θέλω επίση και να υπογραμμίσω την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο παρελθόν ήταν σαν το σαν το πλατωνικό σπήλαιο έβλεπε μέσα από τις σκιές αυτά τα οποία έκανε η Κομισιόν. Ενώ κανείς δεν κοιτούσε πώς λειτουργούσε το ελεκτικό συνέδριο και το ελεκτικό συνέδριο απασχολείται με τις σκιές του στίχους της σπηλιάς. Έχει κάνει κάποιες προτάσεις σε σχέση με τους κανόνες συμμετοχής στα προγράμματα, αλλά και η Κομισιόν είχε κάνει μια προσπάθεια να καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε το ελεκτικό συνέδριο τότε. Είναι λοιπόν απαραίτητο για το επόμενο πρόγραμμα να υπάρξει μια ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και θα θέλω να σας θέσω ένα παράδειγμα. Η απλοποίηση των διαδικασιών στον <clears throat> ορίζοντα 2020 θα πρέπει να σημάνει και μια μεγαλύτερη ε, ανάληψη ευθύνης της Κομισιόν ώστε να γίνεται πιο εύκολα η χρηματοδότηση. Ε, μα ο στόχος δεν είναι αυτό το οποίο θέλει η Κομισιόν να μην έχει προβλήματα με τον έλεγχο του προϋπολογισμού ή με το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν μπορούν να αποφασίζονται οι διαδικασίες με, αυτό το λογικό, με αυτή τη λογική. Όπως είπατε πρέπει να πριτανεύσει και η κοινή λογική κάποια φορά. Λοιπόν, σε συγκεκριμένο επίπεδο είναι χρήσιμο να συζητούμε και για τα διάφορα υποδείγματα ε, κόστους και να εφαρμόσουμε ορισμένε φορές το αγγλοσαξονικό μοντέλο της ε, τιμολόγησης. Από συστημική άποψη αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι απίστευτα πολύπλοκο αυτό το σύστημα. το οποίο λειτουργεί με το να ανταμείβει με ένα συγκεκριμένο ποσό μία συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύστημα, αλλά αυτό απέχει πόρο από το συνηθισμένο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης. Την τελευταία φορά λοιπόν είχαμε πάρει ορισμένα στοιχεία για την <clears throat> συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην, ε, στις προσκλήσεις του ορίζοντα 2020. Το θέμα λοιπόν της υπο, ε, μάλλον της ε, περιορισμένης, της ανεπαρκούς υποβολής προτάσεων ή της υπερβολικής υποβολής προτάσεων είναι κάτι που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ακριβό για μια μικρομεσαία επιχείρηση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα χωρίς να έχει τη βεβαιότητα ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα, πρόβλημα μονάχα υπολογισμών. Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων είναι πολύ πολυδάπανο να είναι κανείς στο πρόγραμμα αυτό, αλλά ανεξάρτητα και από αυτό είναι ήδη πολύ ακριβό <clears throat> να συμμετέχει κανείς στο πρόγραμμα. Δεν έχει νόημα να κοστίζει το 1 τρίτο της επιδότησης που παίρνει κάποιος όταν συμμετέχει στο πρόγραμμα, το 1 τρίτο από αυτό το ποσό να δαπανάται για να μπορέσει καταρχήν να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν είναι βιώσιμο. Επίσης, <clears throat> όταν έχουμε τα λογιστικά συστήματα, όταν για παρόμοια προγράμματα, επομένω για αντίστοιχε ε, παροχέ υπηρεσιών έχουμε τρία διαφορετικά λογιστικά συστήματα, αυτό είναι προγραμματικό. Δηλαδή, αλλιώς καταγράφουν λογιστικά τα πράγματα που κάνουν οι επιχειρήσεις στο εθνικό επίπεδο από ό,τι στο ευρωπαϊκό. Αυτό έχει λογική. Αλλά δεν μπορούμε για παρόμοια προγράμματα να έχουμε διαφορετικά λογιστικά συστήματα. Και ερχόμαστε σε ένα ουσιαστικό θέμα. Είναι σημαντικό για δύο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη να έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο λογιστικής καταγραφής στα εθνικά κράτη που δεν είναι καν αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, πρέπει να έχουμε ένα δικό μας ευρωπαϊκό τρόπο λογιστικής καταγραφής. Μπορεί λοιπόν να γίνεται επομένως <clears throat> το λογιστικό σύστημα της Φιλανδίας να είναι πιο ευνοϊκό για μια φιλανδική εταιρεία από ό,τι θα ήταν αντίστοιχα στην Γερμανία. Αλλά αυτό, αυτές οι διαφορές θα έπρεπε να διατηρηθούν ή θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε κάποιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ότι για τα ίδια σχέδια οι ίδιοι φορείς θα έχουν την ίδια λογιστική καταγραφή. Αλλά σας λέω και πάλι έχει νόημα να έχουμε δύο συστήματα αξίζει τον κόπο να έχουμε εμπιστοσύνη στα εθνικά συστήματα ή πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θέσουμε κάθε φορά που θέλουμε να προχωρήσουμε στην απλοποίηση. Αλλά όταν βλέπουμε τα έγγραφα που έχει παραγάγει η Κομισιόν για τα θέματα αυτά του ελέγχου είναι χιλιάδες σελίδες, τότε δεν έχει κανένα νόημα η απλοποίηση. Ουσιαστικά υπάρχει μια αυξανόμενη πολυπλοκοποίηση και επομένω πρέπει να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο θέμα αυτό. Αν έχει νόημα να έχουμε διαφορετικά συστήματα λογιστική καταγραφή στα εθνικά κράτη από ό,τι στο Κοινοβούλιο, και εγώ μπορώ να σα πω από προσωπική άποψη, θυμάμαι μαζί με τον κύριο Μπούζεκ έχουμε αντιμετωπίσει το πρόγραμμα πλαίσιο 6, το πρόγραμμα πλαίσιο 7, το Horizon 2020. Είχαμε και στο παρελθόν αυτές τις συζητήσεις, γι' αυτό είναι απαραίτητο πρωτού ε, θεσπίσουμε τους νέους κανόνες συμμετοχής στα ερευνητικά πρόγραμμα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να μην μιλάμε για απλοποίηση όταν χρειάζονται 700 σελίδες για να μας εξηγήσουν σε τι συνίσταται αυτή η απλοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απροσδόκητο το συμπέρασμα. Αλλά πιθανότατα αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Επόμενος ο συνάδελφος Σον Κέλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ομιλητή για τη σαφήνειά του και τα διάφορα θέματα. Είπε ότι κάποιοι δικαιούχοι δεν συμμορφούνται λόγω ελλείψους γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Και πιο ανησυχητικό είναι ότι είπε ότι κάποιοι δεν συμμορφωνόταν γιατί δεν ήθελαν να αποδώσουν όπως έπρεπε. Και χρειαζόταν πίεση. Θα ήθελα να γνωρίζω αυτοί που δεν αποδίδουν σωστά. Το κάνουν για πρώτη φορά ε, ή κατά εξακολούθηση. Και αν ναι, ποια δράση έχει ακολουθηθεί εναντίον τους κατά παρελθόν. Και αν επανειλημμένα δεν αποδίδουν σωστά, ε, τι μέτρα θα ήθελε να εφαρμοστούν εναντίον τους. Όλοι πηγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, σε αυτούς, σε διάφορους φορείς, που σκοπίμως εξαπατούν και τελικά ξεφεύγουν. Αυτό αποτελεί προσβολή. Και είναι και απαράδεκτη συμπεριφορά εξάλλου. Δεν άκουσα ποτέ να χρησιμοποιεί τόσο συχνά κοινή λογική εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευπρόσδεκτο αυτό. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Έιλερ, ο συνάδελφός μου, που είπε ότι τρία διαφορετικά λογιστικά συστήματα εφαρμόζονται. Αυτό δεν μου φαίνεται ότι ακολουθεί την κοινή λογική. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν Πού θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την κοινή λογική, σε ποιου τομεί θα μπορούσε να εφαρμοστεί και δεν εφαρμόζεται. Το παράδειγμα του κυρίου Νιέλ ήταν ένα, αλλά δεν έχει νόημα να κουβεντιάζουμε. Αυτό δεν συνέβη για μία βραδιά και μόνο, επί μακρόν χρονικό διάστημα. Άρα είναι και η ώρα προς δράση. Και να σταματήσουμε τα λόγια και να κινηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφε, λέει ο κ. Μπούζεκ. Ο κ. Κοχλιτσέκ έχει το λόγο. Α, η κυρία Κουντρίτσκα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν είναι το ίδιο. Κύριος Κοχλίτσεκ και κυρία Κουντρίτσκα δεν είναι ταυτόσημα. Κανένα πρόβλημα, λέει η κυρία Κουντρίτσκα. Θα μιλήσω πολωνιστή. Λοιπόν, Νομίζω ότι χρειάζεται κάποια καινοτόμα προσέγγιση. Να έχουμε καινοτόμες ε, διαδικασίες ελέγχου. Αυτό είναι σημαντικό. Πιο σημαντικό όμως είναι να δούμε ότι υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες δράσεις που θα το πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφερθήκατε σε απλούστευση. Αυτή την ε- απλούστευση θέλουμε να πετύχουμε. Αν, λοιπόν, αν λοιπόν μια σύμβαση ε, αποτελείται από 700 σελίδες, ένα συμβόλαιο για χορηγία, μια συμφωνία για χορηγία αποτελείται από 700 σελίδες, τότε Είναι περίπλοκα τα πράγματα. Μπορεί να αποκτήσει κανείς αυτά τα χρήματα μόνο αν είναι εμπειρογνώμων ή κάποιος εμπειρογνώμων εξετάσει το έγγραφο. Ή εταιρείε εμπειρογνωμόνων. Και βγάζουν πολλά χρήματα οι εταιρείε αυτού του είδους ε, έτσι. Αυτό σημαίνει δαπάνες, μεγάλες δαπάνες από πλευράς φορέων ερευνητικών για την προετοιμασία κάποιου έργου, κάποιου προγράμματος, κάποιες έρευνας. Οπότε πολύ συχνά οι τυπικές διαδικασίες είναι ο σημαντικότερος λόγος για την ε, απόρριψη ενός αιτήματο για χρηματοδότηση. Έχετε ελέγξει λοιπόν σε πόσες ε, περιπτώσεις έχουν απορριφθεί αιτήσει για χρήματα λόγω, ε, για λόγους τυπικούς. Διότι εν τη αυτή περιπτώση η αριστεία ή η, η επιστημανική ποιότητα ε, που χαρακτηρίζει το αίτημα έχουν μικρότερη σημασία από τη τυπική διαδικασία και τα τυπικά η ε, συμμόρφωση με τυπικές προδιαγραφές. Έχετε λοιπόν τέτοιες πληροφορίες για τυπικούς λόγους πόσες ε, αιτήσει έχουν ε, απορριφθεί. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Ορίστε. Η κυρία Μπίρινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσει. Έχω κάποιες ερωτήσεις, λέει η κυρία Βέρινγκ. Λέει η ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ένα σύστημα ενθάρρυνσης και εντοπισμού συμπράξεων Ευρωπαϊκών Διευθυντικών και Επενδυτικών Ταμείων και του ορίζοντα 2020. Όμως, η πρώτη έκθεση για τον ορίζοντα 2020 περιέχει ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά αυτές τις συνεργασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε λεπτομερή αξιολόγηση του συντονισμού των ταμείων στα πλαίσια της ενδιάμεσης εκθέσεως για τον ορίζοντα 2020 που θα δημοσιευτεί το 2018 φρονείτε ότι αυτή θα, αυτή θα έχουμε επαρκή χρόνο να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα, κενά και συνέπειες μεταξύ. Μετά στο κεφάλαιο 4 της εκθέσεως αναφέρεστε στο επίπεδο σφαλμάτων 4,4% όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ε, συναλλαγές. Ποιο είναι το επιτυχές ποσοστό ανάκτησης των αχρεωστήτων καταφύντων ποσών. Ισχύει για όλα τα ταμεία και μπορεί να είναι αυστηρότερο εκ των υστέρων, ε, μίσος ε, έλεγχος θα μειώσει το πρόβλημα. Υπάρχει ο κίνδυνος καταβολή ε, καταβολής τέτοιων χρηστήτων ποσών και στον ορίζοντα 2020 παρόλο που η διαδικασία των ορίζοντα 2020 είναι απλούστερη. Η έκθεση αναφέρει ότι οι διάφοροι εφαρμοστικοί φορείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά το να καταλήξει κοινή θέση για την εκτέλεση των συστάσεων του ελέγχου για την ανάκτηση ε, των παρατύπων δαπανών. Ποιο είναι το επίπεδο διαφωνίας μεταξύ των φορέων και πώς τελικά μπορούμε να πετύχουμε μια συνέπεια στον αφορά στις προσπάσεις ανάκτησης. Τέλος, η έκθεση καλωσορίζει ένα θετικό βήμα. Δηλαδή, του, κέντρου, Κοινού Κέντρου Υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δαπάνες για έρευνα και καινοτομία για την εφαρμογή των στρατηγικών για τις ε, εκτονιστέρων των ελέγχους του 7ου προγράμματος για την έρευνα και το ορίζοντα 2020. Όμως λέτε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας που διαχειρίζεται πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ του ορίζοντα 2020 επί του παρόντος δεν συμμετέχει στο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το Ινστιτούτο αυτό να ενταχθεί και να ενσωματωθεί στο πλαίσιο ελέγχου και γιατί αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ο κύριος Έλλερ έχει το λόγο. Um, Έχω και άλλες ερωτήσεις όσον αφορά το θέμα. Πώς το ελεγκτικό συνέδριο πραγματοποίησε τους ελέγχους και συνέταξε τις εκθέσεις κατά παρελθόν. Είχε βασιστεί σε κανόνες και στην ε, κατανομή των ποσών. Στην νομική πράξη του ορίζοντα 2020 τονίζεται πολύ περισσότερο ο έλεγχος βάσει αποτελεσμάτων. Ερώτηση σε ποιο βαθμό αυτό ήδη αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί τους ελέγχους, από ό,τι γνωρίζω, το ελεγκτικό σύστημα αυτό καθε αυτό πρακτικά σχετίζεται με το παρελθόν, παραπέμπει στο παρελθόν, ενώ το κομμάτι που βασίζεται από που προέρχεται από την νομική βάση, αντικατοπτρίζεται δομικά από τον τρόπο που επιλέγουμε τους ελεγκτές ή που πραγματοποιούμε τους ελέγχου. Ανοίγεται μια πόρτα για πρώτη φορά στον έλεγχο του EIT γίνεται ο έλεγχος με δύο τρόπους και βάσει του κόστους και σε σχέση και με το αποτέλεσμα ταυτόχρονα. Πώς αντιλαμβάνεστε λοιπόν στην ενδιάμεση έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον ορίζοντα 2020 να το προσεγγίσετε το θέμα. Μπορούμε να παράγουμε στοιχεία που ίσως χρειαστείτε για να συμμορφωθείτε με την νομική πράξη. Επιπλέον. Άλλη ερώτηση. Υπήρχαν κανόνες κατά παρελθόν για τη συμμετοχή. Ήθελαν να δομήσουν κατά κάποιο τρόπο τους λογιστικούς ελέγχους, οι κανόνες αυτοί, αλλά να πλαισιώσουν και την έρευνα, τη χρηματοδότηση της έρευνας. Το κόστος συσχετιζόταν με τις υποδομές τις ερευνητικές και το πόροι κατά πρόγραμμα. Ετίθεται το θέμα επανεπενδύσεων των ποσών δεν το σωστά. Θέλαμε να διαβρύνουμε το πεδίο κάλυψης. Κατά παρελθόν θέλαμε να κινηθούμε απλούστερα, να δίνονται κατά αποκομήν ε, ποσά για τα λειτουργικά έξοδα κλπ. Ερώτηση λοιπόν, οι κανόνες για ένα πρόγραμμα οργανώνουν το, τη σωστή απορρόφηση των χρημάτων και τη δαπάνη αυτών, να μην υπάρχει κατάχρηση ή σχετίζεται ο έλεγχος και με τα αποτελέσματα. Είναι ένα θέμα αρχής που θα πρέπει να απαντηθεί πριν θεσπίσουμε ένα νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και κανόνες συμμετοχής. Ευχαριστώ, ρε Πρόεδρος. Μπορώ να σταθώ, αν θέλετε, σε ένα ερώτημα που θέσατε προηγουμένως και θα ήθελα να το διατυπώσω ίσως με πιο πολύ ακρίβεια για την ποιότητα της διαχείρισης στα σχέδιά μας. Γιατί κάποια από αυτά τα σχέδια την χάνουν διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ορίζοντα 2020 ή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ενώ κάποια άλλα τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, μπορεί να είναι το ίδιο αντικείμενο ή παρόμοιο αντικείμενο σε αυτές τις περιπτώσεις. Βρήκατε κάποια διαφορά σε ό,τι αφορά την, ε, τα αποτελέσματα της διαχείρισης. Πού βλέπετε να υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά από την αποτελεσματικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 100 μελών. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της DG Grow, ο κύριος Patrick Child, να λάβει το λόγο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι αναπληρωτή γενικός Διευθυντή στην ε, DG Grow στο τμήμα έρευνα και ανάπτυξη. Χαίρομαι για την ευκαιρία αυτή να μπορέσω να συμβάλλω στι συζητήσει σα και θέλω να σας, ε, να σας συγχαρώ για την οργάνωση αυτή τη τόσο σημαντική και επίκαιρη συζήτηση θάρρος μας δίνει ότι μια επιτροπή όπως η δική σας ενδιαφέρεται και στα θέματα του οικονομικού ελέγχου σε σχέση με, την, ε, με τον έλεγχο των ΣΥΡΕ. Μα έχουμε ένα χωριστό γενικό ε, διευθυντή που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Είμαστε η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης. Αλλά βοηθούμε και τον πρόεδρο Γιούνκερ στην ανάπτυξη και την απασχόληση και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση αυτή. Να σας πω λοιπόν ότι καταρχήν εμείς έχουμε συνεργαστεί του κ. Μπερενίκ Μέιερ και το ελεκτικό συνέδριο <clears throat> και χαιρόμαστε πολύ για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Βρίσκουμε ιδιαίτερα ότι το κεφάλαιο 5 που είναι το επίκεντρο αυτής της συζήτησης δίνει μια εξισορροπημένη περιγραφή των βελτιώσεων που έχουν γίνει εν ώψη της απλοποίησης των διαδικασιών του ορίζοντα 2020 σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και επίσης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου υποστήριξης που συνενώνει για όλες τις υπηρεσίες, του αποκεντρωμένους φορείς, τις γενικές διευθύνσεις, ένα κοινό χώρο ε, για κατανόηση, για αμοιβαία κατανόηση και με τον τρόπο αυτό έχουμε αυξήσει και τη συνεκτικότητα και έχουμε αυξήσει και την πρόσβαση με νέα πληροφορικά συστήματα. Χαιρετίζουμε λοιπόν τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου και κατανοούμε και αποδεχόμαστε την ε, σύσταση να συνεργαστούμε καλύτερα και με το ελεκτικό συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Η σημερινή συζήτηση νομίζω ότι έχει υπογραμμίσει δύο πολύ σημαντικά θέματα. Πρώτο, την ανάγκη να προχωρήσουμε περισσότερο με την απλοποίηση. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Επιτρόπου Μουέντος Και επίσης έφτασα σχετικά πρόσφατα σε αυτή την Γενική Διεύθυνση και εγώ έχω εντυπωσιαστεί από την πολυπλοκότητα των κανόνων μας. Το το υπόδειγμα για την χορήγηση με τις 700 σελίδες. Περιλαμβάνει και πολλές εξηγήσεις γιατί το αρχικό κείμενο είναι πολύ πιο περιορισμένο σε όγκο. Αλλά δίνουμε εκεί πέρα μια πλήρη τεκμηρίωση. Αλλά οι λεπτομέρειες που έχει το έγγραφο αυτό δεν είναι γιατί εμείς τη βρίσκουμε με τις λεπτομέρειες και τα πιο μακροσκελή έγγραφα, αλλά γιατί όταν ανακύπτουν ερωτήματα και προβλήματα από τους δικαιούχους ή από άλλους εμπλεκόμενους, Προσπαθούμε να δώσουμε σαφείς απαντήσεις και καλή κατεύθυνση ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ενδιαφερόμενοι πώς εφαρμόζονται οι κανόνες μας. Αλλά είμαι και ο πρώτος να παραδεχτώ ότι αν μπορούσαμε να βρούμε απλούστερους τρόπους στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για τους κανόνες συμμετοχής, αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε και να το εφαρμόσουμε δραστήρια. Ένα δεύτερο και εξίσου σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η εξισορρόπηση της έμφασης που έχουμε στο να βλέπουμε τις εισρωές και τις διαδικασίες των, ε, της διαχείρισης των χορηγήσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Σας υπενθυμίζω λοιπόν και την πρωτοβουλία της κυρίας Γεώργεβας μαζί με τον Επίτροπο Μουέτος σε ό,τι αφορά τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για ένα προϋπολογισμό ο οποίος εστιάζει στα αποτελέσματα. Και το πραγματικό ερώτημα είναι εμείς εργαζόμενοι με όλους τους εμπλεκόμενου τους λογιστές, τους αναλογιστές, τους υπολογιστές, το ελεκτικό συνέδριο, μπορούμε να βρούμε ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο να καταμετρήσουμε την επιτυχία των εκροών, των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων μας και όχι μία όλο περισσότερο σε βάθος και ε, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα επαχθή διαδικασία ελέγχου των εισρώων και της διαχείρισης. Νομίζω ότι η εφετινή έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου τονίζει ότι τα ποσοστά ασφαλμάτων που διακριβώνουν για προγράμματα τα οποία βασίζονται σε ε, μια ε, καταποκοπή ε, παροχή κονδυλίων για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, εκεί είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά ασφάλματος από ότι στο παραδοσιακό σύστημα που μετράμε τις εισρωές και την διαχείριση. Αν μπορούμε λοιπόν να κοιμηθούμε περισσότερο προ την κατεύθυνση αυτή μαζί με την Επιτροπή, αυτή μαζί με την Επιτροπή Ελεκτού Προπολογισμού, τότε θα κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Νιώθω απίστευτο ενθουσιασμό για την προσέγγιση αυτή. Για να απαντήσω και μερικά ακόμα ερωτήματα τα οποία τέθηκα. Πρώτα, από όλα για το θέμα των παραλλήλων συστημάτων λογιστική συμφωνώ απόλυτα. Όσο περισσότερο μπορούμε να επιτρέψουμε στου δικαιούχου να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά ή τα εθνικά του συστήματα, τόσο το βέλτιο. Κινούμεθα προ την κατεύθυνση αυτή. Υπήρξε και μια έρευνα μεταξύ των συμμετεχόντων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων κτλ. Όπου πάρα πολλοί δικαιούχοι τώρα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα δικά του συστήματα, τα εθνικά του συστήματα. Εμεί θέλουμε να πετύχουμε εκεί περαιτέρω τροποποιήσει για του εφαρμοστικού κανόνε οι οποίοι θα μα οδηγούσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Έλερ ότι αυτό είναι ένα σωστό δρόμο και αποτελεί και ένα τμήμα αυτή τη κοινή λογική που λέει και ο κύριο Μπρέιτ Μάιερ. Το άλλο θέμα, το θέμα των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών ταμείων και του ορίζοντα 2020 και των διαφορετικών τρόπων ε, διαχείρισης θέσατε των δάκτυλό σας επί των τύπων των ύλων για την διαχείριση αυτών των χορηγήσεων βάσει του ορίζοντα 2020 που γίνεται με ένα κεντρικό τρόπο από την Κομισιόν, ενώ η λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή των διαφορετικών ταμείων βρίσκεται στα χέρια των τοπικών και περιφερειακών ε, φορέων στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν μας έχει αποτρέψει από το να λειτουργούμε με πολύ ενεργό τρόπο στον τομέα αυτό και ο κύριος Μουέντος μαζί με την κυρία ε, Μπούλτς. Επίσης έχει εξασφαλίσει κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά την έννοια των σφραγίδων αριστείας που χαιρετίζει με τον τρόπο αυτό την επίτευξη των προτύπων που θέλουμε για τη χρηματοδότηση στο ορίζον 2020. Δυστυχώς, ελλείψη χρημάτων και επειδή υπάρχουν πολλέ αιτήσει σε σχέση με τη δυνατότητα χρηματοδότηση δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε όλους αυτούς, αλλά τότε αποδίδεται αυτομάτω η σφραγίδα ε, αριστεία, ώστε να ξέρουν οι διαχειριζόμενοι τα διευθυντικά ταμεία ότι είναι καλό το πρόγραμμα αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο επίση θα λυθεί υπόψη στην ενδιάμεση αναθεώσει για τον ορίζοντα 2020 την οποία επεξεργαζόμαστε με στόχο να προχωρήσουμε έτσι περισσότερο στο επόμενο σχέδιο πλαίσιο, μάλλον πρόγραμμα πλαίσιο για τα θέματα αυτά. Ετέθηκε ένα ερώτημα σε σχέση με το πώς εξασφαλίζουμε την συνεκτικότητα σε ό,τι αφορά τις ανακτήσεις κονδυλίων από διάφορους διατάκτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα και μόνο δικαιούχο και εδώ πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια ισορροπία μεταξύ αφενός της ευθύνη των διατακτών να κάνουν κατά περίπτωση για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων και την, από την άλλη πλευρά ανάγκη μεγαλύτερης κεντροποίησης και συνεκτικότητας θα έλεγα ότι η δημιουργία του κοινού κέντρου υποστήριξης και τι ε, υπηρεσίε λογιστικού ελέγχου εκεί μα βοήθησε να πάμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι είναι κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μα. Αληθεύει εξάλλου το ότι το Ευρωπαϊκό Συνδείο Τεχνολογία δεν καλύπτεται από το κοινό κέντρο υποστήριξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το δικό του οικονομικό έλεγχο και τα συστήματα διαχείριση δημοσιονομικών. Και έγινε γι' αυτό μια χωριστή έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ακολουθεί τους ε, κανόνες και υπάρχει η σωστή παρακολούθησή του. Νομίζω ότι κάλυψα πολλά από τα ερωτήματα τα οποία τέρκαν στη συζήτηση. Μόνο το ερώτημα του κύριου Κέλλη. Τι να κάνουμε όταν υπάρχει η θελημένη παραβίαση των κανόνων και κατά και επανάληψη Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική μηδενική ανοχής για τις απάτες. Ο κ. Πέννεμαερ ανέφερε σε περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο στην Όλαφ και εμεί παραπέμπουν αυτά τα ζητήματα στην Όλαφ αν υπάρχουν υποψίες που προκύπτουν από τις δικές μας λογιστικές έρευνε. και παρακολουθούμε πάρα πολύ εντελεχώς τις έρευνες της Όλαφ και αν υπάρξουν ενδείξεις ότι υπάρχουν παραβιάσεις και καταχρήσεις, τα θέματα αυτά παραπέμπονται στα εθνικά, στι εθνικέ αρχές για να λάβουν δράση εναντίον αυτή τη συμπεριφορά. και όπω ξέρουν οι συνάδελφοι, η Κομισιόν έχει ένα σύστημα βάσει του οποίου αυτοί οι οποίοι δεν ακολουθούν τους κανόνες μας ή θελημένα ή προχωρούν σε απάτες μπορούν να αποκλείονται από μελλοντική χρηματοδότηση. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στο να εξασφαλίσουμε ότι η απατηλή ή η κατασυρωή ε, ατασταλής συμπεριφορά κολλάζεται με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο ώστε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να την χάνουν τις πρέπουσες προστασίες και τώρα για τον υπο υπερβολικό αριθμό αιτήσεων και το μικρό ποσοστό επιτυχίας και το μεγάλο διοικητικό άκθος που επιμίζονται αυτοί οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις. αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ και γι' αυτό σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε και έχουμε εισαγάγει την έννοια μιας <clears throat> διαδικασίας δύο σταδίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου στο πρώτο στάδιο παρουσιάζουν οι ενδιαφερόμενοι ένα απλοποιημένο σχέδιο για τις ιδέες τους και έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους δυνητικούς ε, ε, υποβάλλοντες ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθεί το συνολικό άχθος υποβολής. Βέβαια αυτό καθυστερεί τη διαδικασία, αλλά τέτοιες ιδέες σκεφτόμαστε για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, να ζητήσουμε από τον προσκεκλημένο μας να απαντήσει στις ερωτήσεις και τις τελικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζεκ, σας ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Τσάιλτ για τις απαντήσεις του. Δικός μου ρόλος είναι να κρίνω κατά πόσο οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ορθές ή όχι. Και δέχομαι ότι οι απαντήσεις του κύριου Πάντρικ Τσάιλτ κατά την γνώμη μου ήταν περιπορθές. Δεν μπορώ να αποκλίνω. Κάτι το οποίο βέβαια διευκολύνει και το δικό μου το ρόλο. Εγώ θα ασχοληθώ με μερικά ζητήματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που γίνεται και που εκτιμά όλο ιδιαίτερο Γιατί μπορεί να συνεισφέρει σε μια καλύτερη διαχείριση στην έρευνα, στα κονδύλια δηλαδή, της έρευνας και της καινοτομίας. Κύριε Έλερ, είπατε ότι χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, συμφωνώ. Μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες που είναι πολύ ενδιαφέρουσες για την εκπόνηση πολιτικής. Ένα από τα πράγματα που υπογραμμίσατε και ο κύριος Πάτρικ Τσάιλ το ανέφερε είναι η ανάγκη να έχουμε αποτελέσματα τα καταποκοπήν ίσως να είναι μια βελτίωση. Και μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι αν δείτε στο σύστημα αυτό μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό κόστος και το καταποκοπήν. και να υπάρξουν ποσά τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί καλά από το δικαιούχο. Επίσης, σε αυτά που είπατε, ο αξιότιμος Πολωνός ε, συνάδελφος, αλλά δεν τολμώ να επαναλάβω το όνομά σας, μήπως το καταστρέψω με την προφορά μου. Το είπε και ο κύριος Τσάιλτ. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Το να φτιάξουμε μια εικόνα του πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθούμε και το κόστος. Όπως σας είπα πριν, των διαφόρων ε, εταιριών ε, συμβούλων που ετοιμάζουν προγράμματα ε, που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Τσάιλντ επίσης είπε και κάποια πράγματα για την χρήση των εθνικών συστημάτων ελέγχων στο λεκτικό συνέδριο γίνεται συζήτηση για ενιαίες συζητήσεις και ενιαίο έλεγχο. Ο έλεγχος μας για την λειτουργία του EIT, το Κέντρο Τεχνολογίας, του Ινστιτούτο Τεχνολογίας, διαπίστωσα ότι εκεί οι έλεγχοι γίνονται πλήρως και γίνεται ένας, όχι τρεις ή πέντε. Για τον κύριο Κέλλη. Το ζήτημα της επανάληψης, ο κύριος Πάτρικ Τσάιλντ επίσης αναφέρθηκε σε αυτό. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι στο ελεγκτικό συνέδριο καταρτίζουμε τους ελεγκτές μας για να εντοπίζουν πιο συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν την Όλαφ και να ενημερώνουν όχι μόνο την Όλαφ αλλά και, τα, και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές για το τι συμβαίνει στη χώρα τους. Με ρωτήσατε επίσης αν μπορώ να δώσω παραδείγματα κοινή λογικής. Πολύ ωραίο. Ήμουνα δικαστής για πολύ καιρό και ασχολήθηκα με την εφαρμογή των κανόνων. Όντως, είναι επάγγελμα αυτό. Μερικές φορές πιστεύω ότι μπορούν να μάθουν οι ελεγκτές πώς να εφαρμόζουν τους κανόνες και τότε έχουμε την κοινή λογική. Γιατί για να εφαρμόσει ένα κανόνα ξεκινάς από το κείμενο του κανόνα. Αλλά δεν είναι αυτό όλο. Το δεύτερο είναι ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δίνεται ο κανόνας. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό, ποιος είναι ο στόχος του κανόνα. Αν λοιπόν λάβετε υπόψη σας και το κείμενο και το πλαίσιο και τον ε, σκοπό, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε τον κανόνα με κοινή λογική. Για παράδειγμα, το κόστος αυτό των συμβούλων. Εάν ένας δικαιώχος έχει τέτοιο κόστος συμβούλων και πρόκειται για εξωτερικούς συμβούλους, ήταν μια περίπτωση που δεν είχε επιλογή, έπρεπε να ε, πάρει εξωτερικούς συμβούλους, γιατί στη συγκεκριμένη οργάνωση δεν είχαν εσωτερικούς συμβούλους. Ωραία, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Μπορείτε να πείτε, α, παραβιάζετε τους κανόνες γιατί έχετε νοικιάσει εξωτερικούς συμβούλους. Έχετε προσλάβει. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό όμως να μπείτε στη θέση των ανθρώπων που κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά και να καταλάβετε τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Και μετά μπορείτε να δείτε ποιος κάνει απάτη Ποιος απλώς προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αν στον, δημοσιονομικό κανονισμό βάλετε το ότι αν ένας ελεγκτής εντοπίσει σφάλμα είναι υποχρεωμένος να θέσει και ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί έγινε το σφάλμα αυτό και να το γράψει στο χαρτί τότε θα μάθε και γιατί έγινε το σφάλμα και τότε θα βελτιωθεί το σύστημα. Δεν φτάνει το να εντοπίζουμε τα σφάλματα. Ναι, εντάξει, έγινε σφάλμα, ναι. Γιατί όμω, για να μάθουμε. Αυτό θα βοηθούσε πολύ. Και αν πετύχετε να εισαγάγετε έναν τέτοιο κανόνα στον δημοσιονομικό κανονισμό, το ότι δηλαδή ο ελεγκτής έχει την υποχρέωση και οι ελεγκτέ του ελεγκτικού συνεδρίου να αναρωτηθούν γιατί γίνεται το σφάλμα και να επιμείνουν να μάθουν το γιατί, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Έρχομαι τώρα στις πληροφορίες όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και το ελεκτικό πλαίσιο. Αυτό είναι ένα θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υπάρχει και το θέμα των συνεπειών των ανακτήσεων των ποσών. Εδώ ανέφερα κάτι το οποίο προσδιορίζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου εκεί υπάρχει μια αλλαγή, γιατί εμείς σε τήσια βάση δουλεύουμε, ενώ όχι πάντα η Κομισιόν. Οπότε, είναι ενδιαφέρον να δούμε και το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί και αυτό μας δίνει πληροφορίες. Και τέλος, κύριε Έλλερ, στη δεύτερη ερώτησή σας, με ρωτήσατε για την αξιολόγηση για τον ορίζοντα 2020 και την διάμεση αναθεώρηση. Ό,τι έχουμε δει στο PP7 είναι ότι κατά διάρκεια του προγράμματος αλλάζουν οι κανόνες. Και ότι και αυτό ήταν ε, πολύ καλό, δεν βοήθησε και πολύ. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να αξιολογήσουμε τον ορίζοντα 2020, Ποιε θα είναι οι συνέπειε, οπότε η πρότασή μου είναι μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του ορίζοντα 2020 να δούμε αν χρειάζονται και άλλοι κανόνες. Τέλος, για το μοντέλο του πλήρους κόστους μεγάλων υποδομών. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται με προδιαγραφές για να αναγνωρίσει τη σημασία που έχουν οι μεγάλες υποδομές και βάσει αυτών να χρηματοδοτήσει με ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για όλες σας τις παρατήσεις, τις απαντήσεις και πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ετήσια έκθεσή σας. Όντως μας βοηθάει πολύ. Λοιπόν, έχουμε, βλέπετε και μια έκθεση περί εφαρμογής και υλοποίησης για τον ορίζοντα 2020 ε, πώς λειτουργεί το σύστημα, οπότε είναι πολύ καλό που σας ακούσαμε και μπορούμε να συναγάγουμε και κάποια συμπεράσματα από την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα καλέσουμε στην αίθουσα τον κύριο Μοέντος, τον Επίτροπο, να έρθει λίγο νωρίτερα εδώ. Α, ένα λεπτό πιο νωρίς. Ένα λεπτουδάκι. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Commissioner. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε άλλο ένα θέμα μπροστά μας. Υπαριθμών 14 ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την σύμπραξη για καινοτομία και έρευνα στον τομέα, στην περιοχή της Μεσογείου. Ο κ. Κάρος Μουέδας είναι εδώ, Επίτροπος Πέθνος για έρευνα, καινοτομία ε, και τις επιστήμες και αυτό γίνεται στα πλαίσια του διαθρωμένου διαλόγου. Κύριε Επίτροπε, κύριε Μουέδας, που εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να πω ότι κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπείτε και την Πορτογαλία και η Πορτογαλία δεν είναι μεσογειακή χώρα. Δεν είναι, δεν είναι. Έτσι έλεγα κι εγώ. Είναι σημαντικό ερώτημα, σημαντικό ζήτημα βλέπετε, γιατί σας ρώτησα. Διότι στη Βαλτική, στο Συμβούλιο της Βαλτικής, έχουμε και την Ισλανδία. Δεν ξέρω αν η Ισλανδία είναι πολύ κοντά στη Βαλτική θάλασσα, αλλά είναι μέλος του Συμβουλίου αυτού. Και η Νορβηγία και η Νορβηγία τώρα δεν έχει ακτή στη Βαλτική. Κοντά είναι. Η Ισλανδία όμως δεν είναι και τόσο κοντά. Ε, είναι δυνατόν και εσείς λοιπόν να είσαστε μεσογειακή χώρα εκπροσωπώντας την Πορτογαλία. Δεν το αποκλείω αυτό. Είναι σημαντικό το θέμα λοιπόν, συνάδελφοι. Δυνάμει το άρθρο 185 αναλαμβάνουμε αυτή την πρωτοβουλία, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γειτονικές μεσογειακές χώρες επενδύουν σε κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Έρευνας και κοινοτομίας. Είναι η πρώτη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. P2P με άλλα λόγια δημοσι... πρωτοβουλία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που προτάθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια και είναι το πρώτο πρόγραμμα που ανοίχθηκε σε συμμετοχή πολλών τρίτων χωρών. Άρα μπαίνουμε σε νέου τύπου προγράμματα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μας βοηθήσει πολύ στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και χώρες της Βορείου Αφρικής, αραβικές χώρες. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Επίτροπε. Θα θέλαμε να μάθουμε πώς βλέπετε εσείς την όλη α, πρωτοβουλία από πλευρά τη Ευρωπαϊκής επιτροπή και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τα αξιότιμα μέλη που με κάλεσαν να παραστώ εδώ. Με τα χαράς να παρουσιάσω σήμερα την από παλιά αναμενόμενη στατική πρωτοβουλία για την καινοτομία και την έρευνα που καλείται πρίμα. Είναι σύμπραξη για έρευνα και καινοτομία στη Μεσόγειο. Την περιμέναμε διακαώς. Θυμάμαι μάλιστα και είναι ενδιαφέρον που είμαστε πίσω αυτή την αίθουσα. Θυμάμαι λέγω ότι τότε εδώ στην ακρόασή μου, σε αυτή την αίθουσα ήμουνα, καθόμουν εκεί, εκεί κάτω. Και θυμάμαι ότι η κυρία Τόγια, η οποία είναι παρούσα, ο κύριος Μπλάνκο Λόπες ήταν εκεί και ο κύριος Μπορέλη. Και μου έθεσαν μία ερώτηση όσον αφορά την σημασία της πρωτοβουλίας πρίμα και θυμάμαι ότι το Δεκέμβριο του 2014 μόνο, μόλις λίγες μέρες από όταν έβρε καθήκοντά μου σαν επίτροπος διεξήγαμε μία συζήτηση στο Στασβούργο να το πω ξεκάθαρα και σταράτα. Θέλω να προχωρήσω με έναν τρόπο που θα είναι αποτελεσματικότερος για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο, την ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας με άλλα λόγια. Σας υποσχέθηκα να αξιολογήσω προσεκτικά τα πλεονεκτήματα της προτάσεως και μετά να αποφασίσω για την βέλτιστη προσέγγιση. Αυτό ακριβώς υιοθετήθηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων στις 18 Οκτωβρίου που μας πέρασε. Πρώτα απ' όλα θέλαμε στρατηγική σύμπραξη με τους ε, εταίρους μας Νοτιού Μεσογείου για κρίσιμες προκλήσεις. Είναι από τα δύο βασικά θέματα που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Και τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε είναι το νερό και το φαγητό, τα τρόφιμα. Θέλουμε να έχουμε ένα όραμα στην περιοχή ποιε θα είναι οι προκλήσει, τα προβλήματα του μέλλοντο. Μετά, με σημαντικέ οικονομικέ δεσμεύσει που θα αναλάβουν οι χώρες και μετά θέλουμε σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπεται το άρθρο 185 των ε, συνθήκων. Γιατί χρειαζόμαστε την πρίμα. Γιατί ε, υποστηρίξαμε τόσο ένθερμα την πρωτοβουλία. Διότι η πρίμα μέσω έρευνας και καινοτομία στηρίζει τα την επίλυση των μεγαλύτερων προβλημάτων της εποχής μας. Πρώτα απ' όλα, όταν δούμε τι γίνεται με το νερό. Σήμερα 180 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν πρόβλημα ε, όσον αφορά το νερό στη Μεσόγειο. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος, το πρόβλημα της υδροδότησης και λόγω κακής διαχειρίσεως ε, των πόρων και λόγω δημογραφικών αλλαγών. Δεύτερον, κάτι που σχετίζεται με το νερό είναι και τα τρόφιμα. Η γεωργική παραγωγή εξαρτάται πολύ από το νερό. Ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων, άρα είναι στατική σημασία για τη Μεσόγειο και για την απασχόληση και για την διαβίωση του ντόπιου πληθυσμού, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για ανάπτυξη. Τρίτον, πέρα από τα τρόφιμα και το νερό έχουμε και το θέμα της μετανάστευσης. Η μετανάστευση, η έλλειψη καλού συστήματος διαχείρισης των υδάτων και συνέπειε που έχει αυτό για την παραγωγή τροφίμων στην περιοχή δημιουργεί οικονομική και κοινωνική ένταση. Αυτά είναι βασικά αίτια για να μεταναστεύσουν οι άνθρωποι και εντό συνόρων και εκτό συνόρων. Έρευνα και καινοτομία λοιπόν έχουν μεγάλε δυνατότητε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε όμω μια πολύ συντονισμένη προσέγγιση και αύξηση των επενδύσεων για να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε τι λύσει. Λοιπόν, ποια είναι τα προσδοκόμενα ωφέλη από αυτά που κάνουμε. Κρίσιμο ερώτημα αυτό για όλου μα πιστεύω. Χάρη στην κοινή ανάληψη υποχρεώσεων και χωρών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των χωρών τη Μεσογείου στο πρίμα θα δείξει πως η έρευνα μπορεί να μετωπίσει κοινά προβλήματα συναθρίζοντας εμπλεκόμενους φορείς και χρησιμοποιώντας εθνικούς προπολογισμούς. Σημαντικός ρόλος της πρίμα. Να εντάξει λοιπόν εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Σημαντικό κομμάτι αυτό. Τι ούτω τρόπος αποτελεσματικά μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτόμες λύσεις για βιωσιμότητα και διαχείριση, το, σωστή διαχείριση των υδάτων και των τροφίμων. Το πρίμα δίνει έξοχες δυνατότητε ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και οι δημόσιε επενδύσεις θα στηρίξουν επίσης και ιδιωτικέ επενδύσεις. Άρα έχουμε οικονομικά ωφέλη. Όμως θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα και όσον αφορά το περιβάλλον. Και θα βοηθήσουμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις, αυξάνοντα τη διάθεση υδάτων και αντιμετωπίζοντα την αλλαγή του κλίματο. Έτσι θα προσαρμοστούν οι περιοχές στις αλλαγές. Έτσι θα υποστηρίξουμε τον αγροτροφημικό τομέα μέσω καινοτόμων λύσεων για να εξοικονομήσουμε ε, το νερό και να χειριστούμε τα δάφη. Λοιπόν, θα βελτιωθεί η παραγωγή τροφίμων, η διαχείριση των οικοκυριών, θα αυξηθεί έτσι η σταθερότητα στην περιοχή και θα μειωθούν εσωτερικέ και εξωτερικέ πιέσει μεταναστευτικέ. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του πρίμα. Ποια είναι, να σα τα αναφέρω. Ακροθυγός τα σημαντικότερα. Έχει 13, 30, ε, συμμετέχοντες, θα αυξηθεί σε 14. Μου είπαν ότι και η Ορδανία καταφθάνει. Ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει. Νοπάμαντατα, πριν από 5 λεπτά μου το είπαν. Τα 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Έχουμε δύο χώρες συνδεδεμένες με τον ορίζοντα 2020, το Ισραήλ και την Ισία και τρεις χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με τον ορίζοντα 2020, η Αίγυπτος, το, ο Λίβανος και το Μαρόκο. Και τώρα ήρθε και η Ορδανία. Η πρωτοβουλία εξελίσσεται λοιπόν. Η Γερμανία ήδη εξέφρασε επιθυμία να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Η Τσεχική Δημοκρατία επίσης πρόσφατα αποφάσισε να αποσυρθεί λόγω ελλείψεω πόρων μας είπαν όμως ότι ελπίζουν αργότερα να ξαναμπούν. Και η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει το 2018 και θα διαρκέσει 10 χρόνια όσον αφορά τον προπολογισμό του πρίμα. Οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύτηκαν για περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά μέχρι τώρα και 131,5 εκατομμύρια σε είδος. Η Ένωση θα ανταποκριθεί στο ποσό αυτό δίνοντα 200 εκατομμύρια ευρώ. Να τονίσω ότι είχαμε και υποστήριξη του συναδέλφου Επιτρόπου Χόγκαν από την ε, αρχή μας υποστήριζε και θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά την πρίμα. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό του ορίζοντα 2020 και θα έχει σαν στόχο κυρίως στρατηγικά επιλεγμένα πιλωτικά προγράμματα και προγράμματα επιδείξεων. Οι εθνικές οικονομικές συνεισφορές για τις δραστηριότητε αυτές θα γίνουν σε επίπεδα κατάλληλα τεχνολογικά με ανωδική πορεία. Η πρωτοβουλία θα εδράζεται επί στρατηγικού θεματολογίου. Αυτή θα εφαρμοστεί μέσω πολλαπλών διαγωνισμών που θα εφαρμοστούν από διάφορες χώρες. Η υλοποίηση θα, θα ελέγχεται από την ειδική δομική, ε, δομικό φορέα, πρίμα IS. Και θα γίνονται έλεγχοι, εξ των υστέρων επαλήθευση, άρα θα έχουμε ορθή οικονομική διαχείριση λόγω των ελέγχων που διεξάγονται και θα προστατεύονται οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και κάτι άλλο. Το πρίμα είναι ένα κομμάτι του πυλώνα μας. Του πυλώνα για το άνοιγμα στον κόσμο. Είναι προτεραιότητα πολιτικής. Είναι ένα καλό παράδειγμα πώς οδηγεί σε διεθνή συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων. Το πρίμα αυθυγραμμίζεται με μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και κυρίως με την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική πολιτική ασφαλής Ευρωπαϊκής Ενώσεως που παραδέχεται τη σημασία βιώσιμων απαντήσεων για την παραγωγή τροφίμων και τη χρήση των υδάτων και της ενέργειας μέσω αναπτύξεως, διπλωματίας και επιστημονικής συνεργασίας σχετικά με αυτό. Πρέπει να πω ότι πριν μερικέ εβδομάδε, στι 13 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δεύτερη έκθεση προόδου για την εφαρμογή τη ανλόγου στρατηγική. Η έκθεση δείχνει ότι ένα άνοιγμα προ τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, ούτω ώστε να προχωρήσει και να είναι στην πρώτη θέση όσον αφορά τι επιστήμε και τεχνολογία και να δημιουργεί θέσει απασχόληση. Η έκθεση επίση τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν παγκόσμια προβλήματα κοινωνικά μαζί με τρίτες χώρες ευθυγραμμίζοντας θεματολόγια και αυξάνοντας τα αποτελέσματα των προσπαθειών επίλυση προβλημάτων όπως είναι η υγεία και η αλλαγή του κλίματος. Το να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο είναι κάτι που διευκολύνεται να έχουμε κατάλληλο πλαίσιο που διευκολύνει την συνεργασία με ισότιμους όρους για τους ερευνητέ από όλο τον πλανήτη. Σε ένα παγκόσμιο ερευνητικό τομέα, οι ερευνητέ, η επιστημονική γνώση και η τεχνολογία θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τέλος, η έκθεση τονίζει το πώς η στρατηγική δίνει αποτελέσματα όσον αφορά την παγκόσμια στρατηγική για την ε, ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Παραδείγματο χάρη στην έρευνα για τη Αρκτική χρησιμοποιείται επιστήμη για κοινή κατανόηση και για κοινέ λύσεις και για ειρηνική συνεργασία και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Όπως και για το πρίμα, όπως και εγώ έδωσα αυτά αναμενόμενο σε αυτό το πρίμα, περιμένω και από εσά να κινηθείτε καταλήρως ώστε η πρωτοβουλία να εγκριθεί τάχιστα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της α, Θα προσπαθήσω εγώ να διευκολύνω τις συνομιλίε συνομιλίες και να ανακουφίσω τις ανησυχίες και του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό θα είναι σημαντικό για να λειτουργήσει σωστά η σύμπραξη και να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2018 και να δίνει αποτελέσματα, διότι έχουμε και φιλόδοξους στόχους άλλωστε σε συνεργασία με τους μεσογειακούς εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ήταν πάρα πολύ σαφής η παρουσίασή σας για τις δυνατότητες αυτές συμμετοχή των κατών μελών μας σε αυτή τη δραστηριότητα και κατανοώ ότι η πλήρης εκκίνηση του προγράμματος αυτού θα γίνει σε ένα χρόνο περίπου. Ωραία. Πηγαίνω τώρα στον κατάλογο των ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Έλερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Το Κοινοβούλιο είναι ελεκτικός φορέας και θέλει να δει ότι υπάρχει σωστή δαπάνη κονδυλίων, αλλά είναι και ένα όργανο το οποίο θέλει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή εδώ και εδώ υπάρχει υποστήριξη του Κοινοβουλίου και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διευρύνουμε και το ε, εύρος αυτής της πρωτοβουλίας για πολλαπλούς λόγους. Έχει νόημα οικονομικά γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τη Γερμανία, την Μεσόγειο συγγνώμη. Δεν θέλουμε να είναι η Μεσόγειος ένα νεκροταφείο προσφύγων και μεταναστών δεν είναι μια σωστή προσέγγιση. Ίσως και οι πρόσθετε, πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο σημαντικός παίκτη στην περιοχή της Μεσογείου και κοιτάζοντας και την ε, ακτή της Βόρειας Αφρικής, την, Μεσό, την Αίγυπτο, τη Συρία, την ε, Αίγυπτο. Έχουμε μόνο δύο ερωτήματα να σα θέσω. Πρώτα απ' όλα, αναφερθήκατε ως ένα πυλώνα το θέμα της τροφιμικής ασφάλειας, της παροχής τροφίμων. Και εδώ θα έπρεπε ίσως να σκεφτούμε και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και τις αρμοδιότητες του στον τομέα αυτό θα μπορούσε να δώσουμε μια νέα όθηση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο έχει διατυπωθεί και υπήρξε και θέληση των μεσογειακών χωρών να χρησιμοποιήσουν αυτή την πρωτοβουλία και να ενισχύσουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι σε μεγάλο βαθμό η... ο κανονισμός αυτού του Ιδρύματος σε μεγάλο βαθμό οδηγήθηκε και από τους συναδέλφους της Μεσογείου. Και έχουμε εξάλλου και μία περαιτέρω πλειάδα θεμάτων στα οποία θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, όπως είναι η ευφυής e e πόλη. Μπορούμε λοιπόν με τέτοιες ε, οθήσεις να πείσουμε το Ινστιτούτο αυτό να ασχοληθεί και με ευρύτερες πρωτοβουλίες που εντάσσονται στον ορίζοντα 2020. Θα ήθελα να έχω λοιπόν την άποψή σας για τα θέματα αυτά και επίσης έχουμε και την ιδέα επίσης ότι εφόσον μιλάμε για το ευρύτερο πλαίσιο της ασφάλειας, θα ήταν μια ευκαιρία να δούμε λιγάκι περισσότερο και τα θέματα ασφάλειας μέσα στον ορίζοντα 20 που έχει να κάνει και με τις σχέσεις της ε, πρωτοβουλίας αυτής της έρευνας για τις πολιτικές πτυχές της ΚΕΠΑ, γιατί και η Μεσόγειος είναι ένας χώρος που υπάρχουν πολλές ανησυχίες για τα θέματα ασφάλειας. Ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσατε να ασχοληθείτε λιγάκι και με, τις, με τα καθήκοντα αυτά τα οποία αφορούν τις ανάγκες πολιτικ... έρευνας για την πολιτική πτυχή των αποστολών και ΕΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόγια από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε για τη μνήμη που έχετε που αποδείξατε ότι έχετε σήμερα, που σημαίνει ότι δίνετε μεγάλη προσοχή στο Κοινοβούλιο και ευχαριστούμε γι' αυτό. Η παρουσίασή σας, όπως είπε και ο πρόεδρος Μπούζεκ, ήταν ιδιαίτερα σαφής. Λοιπόν, έχουμε πλησιώσει πολύ κατά πράγματα. Από εν συντομία, όχι μόνο ενδιαφερόμενες χώρες εν πρώτης, όλοι ενδιαφερόμαστε, διότι η ανάπτυξη Μεσογείου πιστεύουμε ότι είναι κάτι καλό για όλη την Ευρώπη και τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή μας θέση εκεί σε αυτό το σημείο του κόσμου. Και είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους μας. Αν και σήμερα ε, είναι παρούσε περισσότερο οι ενδιαφερόμενες χώρες και η Γερμανία συμπεριλαμβάνεται και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι κινητήρας ανάπτυξης η έρευνα, οικονομικής, κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης. Πιστεύω ότι προ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά για να λάβουμε υπόψη τις πάρα πολλέ προσδοκίες που υπάρχουν στις χώρες του Νότου. Έχουμε σαφές νομοθετικό πλαίσιο, αλλά πρέπει πραγματικά να λάβουμε υπόψη τις προσδοκίες που έχει ο κόσμο, διότι αυτό που θα κάνουμε θα γίνει τοπική κληρονομιά, θα γίνει και κτημένο πραγματικά δικό του. Πρέπει να υπάρξει πολύ ε, εντατικό διάλογο. Χαίρομαι για την παρατήρηση που είπατε αυτό όσον αφορά την καινοτομία και το open innovation κλπ. Διότι πιστεύω ότι το είδος της έρευνας, αυτά, αυτή η που αναφέρατε, ε, διευκολύνουν το, το νερό, τα τρόφιμα, η ενέργεια, διευκολύνουν την ανάπτυξη του ανθρώπου. Είναι στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Ε, πρέπει να εργαστούμε επ' αυτόν. Και έρευνα που αφορά την καινοτομία, ε, ανάπτυξη, οδηγεί στην ανάπτυξη των πολύ μικρών και των μικρομεσών επιχειρήσεων. Είναι παράγοντες ανάπτυξης τοπικής οικονομίας που ξεκινά από την έρευνα. Ε, από που ανέφερε ο συνάδελφος ε, ο κ. Έλλες του ΚΙΚ με την έρευνα για, την, για τα τρόφιμα κλπ. Πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις λοιπόν, κοινέ προσπάθειες. Δεχόμαστε αυτά που είπατε σήμερα. Χρειάζονται θετικές προσεγγίσεις. Έχουμε και το σχέδιο για την Αφρική που, ετοιμάζει, που εξετάζει η Επιτροπή ΔΕΒΕ και η Επιτροπή Ανάπτυξη. Ένα καινούριο ταμείο που δημιουργείται. Υπάρχουν κάποιε σχέσει, είναι διαφορετικά κεφάλαια. Αυτέ οι παρεμβάσει που έχουν στόχο ανάπτυξη δυναμικού των οικονομικών προγραμμάτων ίσω να μπορούν να σχετιστούν και με αυτό το πρόγραμμα. Ίσως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, ε, διότι μιλάμε για δικού μα πόρου ε, και δικά μα αγαθά. Ε, μιλάμε για τους πόρους ε, των μεσογειακών χωρών. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να συναθρήσουμε όλους τους πόρους που διαθέτουμε. Ελπίζω να αρκούν. Ελπίζω να είναι γενναιόδωρος ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για να έχουμε τους αναγκαίους πόρους για να πετύχουμε τους στόχους του φιλόδοξου αυτού προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Βιέρη από την Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Χαιρετίζω την Πορτογαλία. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα σας. Είχα εκεί μια συνάντηση με πανεπιστήμια όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 και την ε, έκθεση εφαρμογή που θα ακολουθήσει. Και έχω μια ερώτηση. Ο... Τα κονδύλια είναι 80 εκατομμύρια για τον ορίζοντα 2020 και συμμετέχουν διάφορα Ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Κάθε Ινστιτούτο όμως, κάθε ερευνητής, κάθε πανεπιστήμιο ζητάει τελικά περισσότερα χρήματα. Έχετε ένα νέο σχέδιο. Ωραία. Υπάρχουν χρήματα, θα κρατήσουν για κάποιο χρόνο, αλλά θα Ξανάρθε η ίδια ερώτηση. Τα πανεπιστήμια, δηλαδή οι ερευνητές, θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα. Πώς θα προσαρμοστείτε, πώς θα το λύσετε αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Μακάρι. Ευχαριστώ κυρία μου για την σαφή σας ερώτηση. Και ο κύριος Κοχ Λιτσέκ τώρα από την Γκουε. Αυτή τη φορά είναι ο ίδιος ο κύριος Κοχ Λιτσέκ, ο του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κάποιος συνάδελφος θέλει να πάρει τη θέση μου πριν από μένα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, στην ηλικία μου πια δεν βιάζομαι. Τέσσερα σχόλια έχω. Ο χώρος της Μεσογείου αντιμετωπίζει το πρόβλημα του νερού που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πρέπει να δημιουργήσουμε φράγματα και πηγάδια και υδατοφράκτες. Οι Τσέχοι έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό σύστημα στη Λιβύη, το οποίο δυστυχώ έχει καταστραφεί τώρα και το Μαρόκο έχει δημιουργήσει φράγματα από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει λοιπόν συσσωρευμένη, συσσωρευμένη εμπειρία για τα θέματα αυτά. Το πρώτο ερώτημα μου είναι λοιπόν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με το σχέδιο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται να έχουν πόσιμο νερό και επίσης νερό για την άρδευση. Η κυβέρνηση στο Μαρόκο έχει ένα σχέδιο υποδομών, αλλά πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και άλλες χώρες για τα θέματα αυτά. Τι θα γίνει με την Αργερία, Η, η Λιβύη ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι η κεντρική κυβέρνηση στη Λιβύη, αλλά για όλες τις χώρες της ε, Μεσογείο υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Ίσως μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Η άδευση και η φύτευση ορισμένων ειδών δασών. Όλα αυτά μπορεί να είναι σημαντικά. Εμείς θέλουμε να έχουμε και φύτευση δασών που θα εμποδίσουν την επέκταση της Σαχάρας προς τα βόρεια. Δεν έχω δει άλλα τέτοια σχέδια, αλλά ξέρω ότι στη Αίγυπτο θα φυτέψουν φοινικοδάσει σε ορισμένε περιοχές με αυτό το στόχο. Θα κάνουμε κάτι σχετικό. Και αυτό είναι σημαντικό και για την Ιορδανία και άλλες χώρες. Και πάλι εμείς ως Τσέχοι είμαστε πολύ πεπειραμένοι στα θέματα αυτά. Σημείο 4. Η προστασία της ε, ε βλάστησης στην Τινησία. Έλαβε χώρα ένα πείραμα όπου προστατεύσαν ορισμένα αγροτεμάχια από τις κατσίκες. Δεν μπορούσαν να πούνε οι κατσίκες εκεί. Και έτσι ξεκίνησε η αποκατάσταση της ε, βλάστησης. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε λοιπόν κάποιες περιοχές από τα εγωπρόβατα και τα βόηδη και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκατάσταση της ε, βλάστησης. Και ένα άλλο θέμα αφορά τη Συρία όπου είναι πολύ σημαντικό και το θέμα των τροφίμων, της παραγωγής τροφίμων. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την κεκτημένη εμπειρία από τη Συρία, η οποία στο παρελθόν μπορούσε να αρδεύει μεγάλες εκτάσεις από τη στιγμή που θα σταθεροποιηθεί λοιπόν η κατάσταση στη Συρία, τι θα κάνουμε για να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν τα σχέδια αυτά. Τέτοιου είδους εμπειρίες λοιπόν πιστεύω μπορούμε να μεταλαμβαδεύσουμε και φυσικά ένα τέτοιο πρόγραμμα όπως το πρίμα θα μπορούσε να προσφέρει τέτοιες δυνατότητες στους εταίρους μας και τις κυβερνήσεις μέσα σε μια συμφωνία συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόχλητσιτς. Ε, κυρία Γκουντλίσκα, έχετε το λόγο. Αυτή τη φορά βρήκα το σωστό όνομα, έχω δίκιο, Λέω ο Ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Κουντρίσκα, Κύριε Επίτροπε, είπαμε ήδη ότι επισκεφθήκαμε την Πορτογαλία και την Ανδαλουσία και πρέπει να πω ότι αναφερθήκατε, αναφερθήκατε στο πολύ καλό αυτό consortium που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση των υδάτων. Επίσης αναφερθήκατε στις ωκεαναγραφικές μελέτες και πρέπει να πω υπάρχει ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Υπάρχουν βέβαια ε, κάποια προβλήματα όσον αφορά τις προδιαγραφές για τα πανεπιστήμια και στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει πολύ ισχυρή βιομηχανία η οποία βιομηχανία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και να χρησιμοποιήσει στην πράξη καινοτόμε ιδέες. Είχε υποθεί στις συζητήσεις λοιπόν με τους εταίρους ότι θα ήταν σημαντικό να παρασχεθούν ε, κίνητρα για τις νεοφυείς ε, επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις παλαιότερες, για να ενδιαφερθούν. Και όσον αφορά το πρίμα, πρέπει να πω θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ποια θα είναι τα ε, χρονικά όρια που θα θέσουμε, το χρονοδιάγραμμα. Πώς θα μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 11 κράτη-μέλη συνεπέραναν ότι οι πόροι ε, πηγαίνουν προς τις ίδιες χώρες και τους ίδιους δικαιούχους και ίσως θα ήταν καλό να γίνει πιο αξιοκρατική διανομή των, των πόρων. Να έχουμε αξιοκρατικά κριτήρια. Θα πρέπει έτσι να γίνει βέλτιστη χρήση των, των πόρων. Αναφερθήκατε και σε κάτι άλλο. Αναφερθήκατε σε διάφορα επίπεδα επιστημονικά και στις αδερφοποίησεις πόλων προσπαθούμε, μάλλον στην αδελφοποίηση και στη συνεργασία των διαφόρων φορέων ε, υπάρχει προσπάθεια να υπάρχει συνεργασία με τους καλύτους επιστήμονες. Πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι θεσμοί στην κοινή αυτή προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί φαινόμενο μόχλευσης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και να φτάσουμε στα βέλτιστα επίπεδα επιστημονικών ερευνών. Αλλά όχι μόνο στην έρευνα, αλλά γενικότερα να κινηθούμε σε πολύ υψηλά ποιοτικά επίπεδα. Πρέπει να έχουμε πολύ ποιοτικά αποτελέσματα. Και να υπάρχει και κάλυψη του κενού που έχουν οι πιο ε, περιοχές. Στην περίπτωση Πορτογαλίας, Ανδαλουσίας, Νοτιού Ισπανίας υπάρχει έλλειψη σωστής δικτύωσης ε, για να μπορούν να διοχετευθούν καλύτερα επιστημονικές δραστηριότητες. Λοιπόν, πρέπει και εμπειρικά να κινηθούμε και όχι μόνο εκτελεστικά. Έχω κάποιες ερωτήσεις. όλες οι έρευνες. Θα έχουν πρακτικό χαρακτήρα. Θα βοηθήσουν να αναπτυχθούν ε, ε, βιομηχανικές υποδομές εκεί που λείπουν. Θα, θα γίνει κάτι να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις. Όσον αφορά τις έρευνες, μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εμπειρία μας και να κινηθούμε και κάπως πιο εμπειρικά. Κυρία Κάμπος Λούις. Ε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον ε, Επίτροπο για την προσπάθειά του τελικά να προχωρήσει το πρίμα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο έργο και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Επίτροπος βοήθησε πάρα πολύ και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε αυτές τις ευχαριστίες. Και εγώ λοιπόν, όπως είπαν και οι περισσότεροι προλαλήσαντες, πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Όχι μόνο για τους λόγους ε, που είπαμε, την ε, γεωργία, το νερό, αναφίβολα, αλλά και γιατί πρόκειται για ένα πολύ βασικό μηχανισμό ανάπτυξης κοινωνικής και οικονομικής και θα βοηθήσει πάρα πολύ και την Νότια Ευρώπη και την Βόρεια Αφρική και είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε και να προχωρήσουμε ώστε να καταστεί επιτυχία. Δύο ανησυχίες, δύο προτάσεις θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, η επιλογή της γεωγραφική δεν έγινε τυχαία. Είναι ότι χρειάζεται λόγω της μετανάστευσης, της οικονομικής ανάπτυξης κλπ. Δηλαδή, η επιλεγμένη περιοχή αποτελεί στοιχείο κλειδί και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή αυτής της περιοχής. Δεύτερον, τα προγράμματα που θα επιλεχθούν είναι αυτά τα οποία έχουν περισσότερη τεχνολογική ανάπτυξη, είναι πιο κοντά στην αγορά. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας τη δυνατότητα που έχουν οι χώρες αυτές όταν θα συμμετέχουν από πλευράς έρευνας και καινοτομίας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή. Και τέλος, είναι σημαντικό η συμμετοχή των χωρών που εγώ χαιρετίζω να συνεισφέρουν οικονομικά. Όχι μόνο τη περιοχή που έχει επιλεχθεί, αλλά και γενικότερα. Είναι ένα βασικό πρόβλημα. Η χρηματοδότηση έπρεπε πρώτα να λυθεί. Οπότε η συμμετοχή των ε, χωρών και αυτών που έχουν δυσκολία και αυτών που δεν συμμετέχουν στην ε, ζώνη την επιλεγμένη πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ τον κύριο που Είναι πολύ θετικό να σας έχουμε πάλι στην Επιτροπή μας. Γιατί θυμάμαι και τη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή αυτή πριν από λίγους μήνες και δείξατε μια μεγάλη δέσμευση για να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία και επομένως είναι πολύ θετική η παρουσία σας και εγώ χαιρετίζω αυτά που είπατε προηγουμένως. Επειδή έχουμε από τη Μάλτα, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό κι είναι η αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, γιατί για μένα η πρωτοβουλία πρίμα είναι κάτι που μπορεί να φέρει κοντά χώρες της Μεσογείου, που είναι μια δύσκολη περιοχή αυτή τη στιγμή, αλλά συγχρόνως μπορεί να ενώσει αυτές τις χώρες, να τις φέρει πιο κοντά μεταξύ τους και να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές μας χώρες στην Μεσόγειο. Χαίρομαι λοιπόν που αναφερθήκατε και στο γεγονός ότι θα εστιάσει εκεί πέρα ιδιαίτερα η πρίμα. Θέλω να υπενθυμίσω αυτά που είπατε, το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και θα θέλω να παρατρύνω όλους τους συναδέλφους μου να ακολουθήσουν ένα πιο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για αυτό το θέμα και υπογραμμίζω ότι η Προεδρία της ε, Μάλτας κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα αυτό στο πρώτο μισό του 17 και χαίρομαι που άκουσα και την κυρία Τόγια να τονίζει την ε, θέλησή της να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό και έτσι να προχωρήσουμε με την πρωτοβουλία πρίμα. Χρειάζομαι όμως κάποιες διευκρινήσεις εκεί από την Κομισιόν, ιδίως για τους δύο πυλώνες, την ε, ε, προσέγγιση του άρθρου 6 για τους δύο πυλώνες θα μπορούσατε να μας εγγυήσετε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα ε, συμμετάσχουν δωρεάν, δηλαδή χώρες του ορίζοντα 2020 θα πρέπει να πληρώνουν και αν θα υπάρξει πρόβλημα να μεταφερθούν κάποια χρήματα στον πυλώνα 2 και ένα άλλο θέμα που θέλω να σας αναφέρω έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πρόταση αυτή ως έχει αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη τεχνολογική ικανότητα. Ενώ οι εθνικές κατά κάποιο τρόπο δραστηριότητε θα εστιάσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τεχνολογίας. Γιατί να μην καλύψει όμως η ευρωπαϊκή συνεισφορά και όλα τα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, ποιες είναι οι απόψεις σας για το θέμα αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Η κυρία Γέρνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε με τον προηγούμενο προσκεκλημένο που είχαμε εδώ, μας μίλησε για τον ορίζοντα 2020 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κονδύλια έρευνας και καινοτομίας. 100 εκατομμύρια πάνε στο πρίμα και 200 προστίθενται από τις διάφορες χώρες. Η ερώτησή μου είναι εξή. Τα κονδύλια πρίμα λοιπόν παραμένουν καινοτομίας και έρευνας κονδύλια ή πρόκειται για νέα κονδύλια διαρθρωτικού τύπου. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Ήταν για την καινοτομία και την έρευνα. Θέλω να ξέρω λοιπόν τι από τα δύο συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ζητά άλλο το λόγο. Θα μπορούσε να είναι και δεύτερη φορά. Όχι. Δεν ζητά άλλο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, για τις συστάσεις, για τη σκληρή δουλειά που έκαναν όλοι για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσω απαντώντας κάθε ερώτηση ξεχωριστά όπω συνήθως κάνω. Ευχαριστώ κυρία Έλλερ, ευχαριστώ Κρίστιαν. Ευχαριστώ για τις δύο ερωτήσεις σου και για αυτά που είπες για τη μετανάστευση και το ρόλο της Ευρώπης, το μελλοντικό ρόλο της Ευρώπης. Πρέπει να είναι ρόλος ανοίγματο. Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το λάβαρο της ε, Ευρώπης. Όσον αφορά αυτό που είπες αρχικά, το ΚΙΚ για τα τρόφιμα, θα μιλήσω με τον συνάδελφο Ναβράσιτς, είναι καλή ιδέα, θα συνομιλήσω με εκείνον με τους συναδέρφους για το γεφύρωμα των νέων μέτρων για τα τρόφιμα και τις πρωτοβουλίες που συζητάμε εδώ. Λογικό. Για το δεύτερο που είπες, για την ασφάλεια. Άκρος ενδιαφέρον και αυτό. Θα γίνει πολλή δουλειά τώρα, εδώ, στο Κοινοβουλίο και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που το πρότεινες. Με τα χαράς να βοηθήσουμε για να συμπεριληφθούν όλα αυτά στην προσπάθειά μας. Ευχαριστώ λοιπόν για τις καλές σου ιδέες. Κυρία Τόγια, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μόνο, βεβαίως, βεβαίως, δεν μόνο. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και να συνομιλούμε για κάτι που σας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Υπογραμμίσατε κάποια σημεία Είπατε να δούμε, για το, να δούμε τι μπορεί να γίνει το νέο στρατηγικό ταμείο για την Αφρική, το νέο ΕΦΣΙ την Αφρική που το εξετάζει συνάδελφο ε, ε, Μογκερίνη και το ΕΦΣΙ 2, αν περιέχει εργαλεία τα οποία περιέχει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ή τα τρόφιμα και το νερό και πώς αλληλοσχετίζονται τα διάφορα διαθέσιμα μέσα και πώς συσχετίζονται με το πρίμα. Αυτά πράγματι είναι σημαντικά που θέσατε. Και το νέο ταμείο ή το νέο σχέδιο Juncker ή το FC2 αυτό το ευρωπαϊκό και αυτό που δημιουργείται για εκτός, ε, χώρες εκτός Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αναφερθήκατε επίσης και στο εξής ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην καινοτομία στον τομέα των τροφίμων και της διαχειρίσεως των υδάτων και η ώρα όπου ο ψηφιακός ε, κόσμος έρχεται σε επαφή με τον κόσμο της διαχειρίσεως των υδάτων και των τροφίμων. Και εδώ το πρίμα θα γεφυρώνει τους διάφορους τομείς. Και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να συσχετίζει τα τρόφιμα με το νερό, και να τα διασυνδέει και με τον ψηφιακό κόσμο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα προχωρήσουμε, λοιπόν. Νομίζω ότι άκουσα δύο ερωτήσεις. της κυρίας από εκεί, κυρίας Βίλια Είπατε ότι επισκεφθήκα την πατρίδα μου. Είπατε ότι θέλετε να σας απαντήσω σε δύο σημεία. Μία ερώτηση αφορούσε τον προπολογισμό και το μέλλον. Είναι δύσκολες οι επιλογές που πρέπει να γίνουν. Χαλεπεί οι καιροί που περιμένουν την Ευρώπη. Μία επιλογή έχουμε έρευνα, καινοτομία και επιστήμες και αριστεία στους τομείς αυτούς. Προτείναμε λοιπόν για τα επόμενα χρόνια 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πολύ καλό για την Ευρώπη. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να, να λάβουμε αποφάσεις πολύ γρήγορα. Θα γίνουν και συζητήσεις στο Κοινοβούλιο που είναι σημαντικότατες και ελπίζω να με βοηθήσετε σε αυτό το σημείο. Μέσω της προτάσεως θέλουμε να προωθήσουμε την αριστεία και να δούμε απ' την άλλη πώς οι χώρες που δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο της αριστείας να αναρριχηθούν στην κλίμακα της αριστείας. Και εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο σας ερώτημα. Ρωτήσατε, αυτό θα φτιάξουμε κάτι παρόμοιο με τα διαθετικά ταμεία. Καταλαβαίνω τι υπονοείτε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο λέμε το εξή. Αν ο βασικό στόχο μα είναι αριστεία, πώ μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνου που έχουν μείνει πίσω να αναρριχηθούν την κλίμακα τη αριστεία. Μεγάλη πρόκληση αυτή. Αν δεν βρούμε λύση θα έχουμε ε, διαφορά μεγάλη. Δείτε τι γίνεται με την παραγωγικότητα σήμερα στην Ευρώπη και την παραγωγικότητα εν γέννη. Τι διαπιστώνετε. είναι στα χέρια των πολύ καλών παραγωγικών εταιριών η παραγωγικότητα, αλλά δεν γίνεται διάχυση της παραγωγικότητας στις εταιρείε που είναι μέσου όρου. Και η παραγωγικότητα είναι στον τομέα μόνο της πληροφορικής. Και πρέπει η παραγωγικότητα να φτάσει στον κόσμο και σε άλλους τομείς, τρόφιμα, νερό, υγεία, ενέργεια. Όλα αυτά σχετίζονται με την αριστεία που είναι κάτι που καλύπτεται τον ορίζοντα 2020. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Διότι με την ερώτησή σας αισθάνθηκα ότι αυτό είχατε κατά νου. Τώρα θα εξετάσουμε και άλλα. Όχι, αριστεία, αριστεία, αριστεία και ξανά μανά αριστεία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους και αυτοί να είναι άριστοι. Μετά, μια άλλη ερώτηση ετέθη του κυρίου Κόλιτσεκ, αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Σημαντικό αυτό που θέσατε. Σημαντικά στοιχεία. Σε κάποια από αυτά που θέσατε θα απαντήσω αργότερα. Μπορείτε να βοηθήσετε και στη διεξαγωγή των συζητήσεων στο Κοινοβούλιο για άλλες χώρες που είναι σημαντικές και πρέπει να τις βοηθήσουμε. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του πρίμα. μαζί με τις χώρες εταίρους μπορούμε να κινηθούμε μαζί, να τις βοηθήσουμε να αναρριχηθούν. Αναφερθήκατε στις εμπειρίες, την εμπειρία που έχετε αποκομίσει από το Μαρόκο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Μαρόκο. Όσον αφορά τη μηχανική έχουν πολύ καλή εμπειρία. Πώς η μηχανική αυτή εμπειρία από τον μηχανολογικό τομέα μπορεί να ταιριάξει με την καινοτομία τώρα που κινούμεθα πιο πολύ προς τον ψηφιακό χώρο. Άρα η καινοτομία των επιστημών και οι εφευρέσεις και η τεχνολογία πρέπει να συνδεθούν με άλλους τομείς ευρωπαϊκούς. Αυτό θα κάνουμε στα πλαίσια του πρίμα. Θα γίνεται σχέσεις με πολλούς ομοτήμους μας σε αυτές τις χώρες, διότι έχουν θύλακες αριστείας εκεί. Έχουν πετύχει πολύ θετικά πράγματα και μπορούμε να συνεργαστούμε. Αν δείτε τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να επιληθούν ε, με κάποια απομονωμένη προσέγγιση μόνο από κοινού. Μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες και συγκεκριμένες απαντήσεις για τη Συρία και για άλλα ερωτήματα που θέσατε αργότερα μαζί με την ομάδα μου. Το πρίμα θα βοηθήσει όλες τις χώρες αυτές, διότι αν προοδεύσεις και αν βρεις καλύτερες λύσεις, όλοι ωφελούνται. Πολύ μεγάλο βήμα βοηθείας προς όλους είναι η πρωτοβουλία μας. Μετά. Η κυρία Γκοτρίκα ε, επισκέφθηκε εκείνη την Πορτογαλία. Ευχαριστώ που το είπατε αυτό. Για την ομαδοποίηση, αδελφοποίηση κλπ. Τις επόμενες δύο εβδομάδες περίπου, εντός σε δύο εβδομάδων, θα σας δώσουμε κάποιες ειδήσει για το teaming και το twinning, για τη δημιουργία ομάδων και αδελφοποίηση. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καλές ειδήσει όσον αφορά διάφορες δράσεις στον τομέα teaming και twinning. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα τώρα. Αλλά παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας επόμενες εβδομάδες. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση την άλλη, να εξετάσουμε το μέλλον, να δούμε τι θα πρέπει να επενδυθεί. Πρέπει να δούμε πώς να βοηθήσουμε τις άλλες χώρες να φτάσουν σε επίπεδα αριστείας και για να γίνουν άριστες οι χώρες, να τις βοηθήσουμε να γίνουν άριστες, είναι κοινή προσπάθεια, δεν είναι τους κάνουμε χάρη, το χρειαζόμαστε. Αν δεν είναι άριστες οι άλλες χώρες, δεν είμαστε και εμείς άριστοι. Εμένα πάντα μου αρέσει να λέω μια ιστορία που μου είπαν προκαιρού, αλλά που μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Ε, κάποιος ο Λούκα Παρμιτάνο μου το είπε αυτό, ένας Ιταλός. Εξηγεί την επιστήμη σαν κανέναν άλλον τα επιστημονικά θέματα. Και συζητούσαμε το θέμα του Τίμινγκ και του twinning. Και μου λέει, κοιτάξτε, σε επιστήμες έχουμε πυραμίδα. Αν θέλεις να βάλεις την κορυφή της πυραμίδας, που είναι η αριστεία, για να βάλεις την κορυφή, μαθηματικά μόνος τρόπος υπάρχει. Να αυξήσεις τη βάση. Να χτίσεις την πυραμίδα, με άλλα λόγια, για να βάλει την κορυφή τη. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε, το έχουμε στην καρδιά μας αυτό, το επιθυμούμε διακαώς και θα κάνουμε τα δέοτα. Έλλειψη της μεγάλης βιομηχανίας, λέει η κυρία Κουντρίσκα. Στην Ανδαλουσία, στο Καδίς και το ίδιο ισχύει και αλλού, σε άλλες χώρες. Δεν έχουμε επαρκή αριστεία. Πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα? Απάντηση. Ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουμε. Όπως το είδε και το Κοινοβούλιο, άλλωστε, όταν σχεδιάζαμε τον ορίζοντα 2020, είναι να συνεργαστούν οι άνθρωποι. Όπως την ομαδοποίηση και στην αδελφοποίηση. Teaming και twinning. Είναι ο μόνος τρόπος. Όταν μαζεύεται ο κόσμος και συνεργάζεται, και συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα στη βιομηχανία ή στα πανεπιστήμια, τότε βελτιώνονται. Και τότε δημιουργείται το συνέστημα της υπερηφάνειας, ότι αν συμμετέχει σε μια ομάδα μπορείς να συμμετέχεις στις εργασίες ενός υπέροχου πανεπιστημίου αυτό δημιουργεί και ένα αίσθημα υπερηφάνεια για την ομάδα που συνδράμει στην αναρρίχηση τη κλίμακα αριστεία Και όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τα αποτελέσματα του εργαλείου τη μικρομεσαία επιχειρήσεις έχουν δείξει ότι κάποιε από τι χώρε που αναρριχώνται στην κλίμακα έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά περισσότερα προγράμματα, όσον αφορά τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το σχετικό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που έχει βοηθήσει τι εταιρείε αυτέ να αναπτυχθούν και να αυξηθούν σε αριθμό σε διάφορε χώρε. Μην σα πω τώρα και για εκείνους που λαμβάνουν τις χορηγίες του εργαλείου αυτού. Πέρσι έδωσα 5.000 δολάρια σε κάποιον από την Κροατία και μου λέει λόγω των χορηγιών μπορώ να είμαι στην Κροατία μπορώ να δημιουργήσω το εργαστήριό μου να εργαστώ στη χώρα και δεν χρειάζεται να είμαι σε άλλη χώρα είπε η ερευνήτρια και έτσι μπόρεσε να δημιουργήσει τις ίδιες τις ευκαιρίες ε, είναι ένα υπέροχο ε, ε, εργαστήριο σε Κροατία που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερεύνας. Ωραία. Τώρα <clears throat> έρχομαι στο τέλος. Πάντα στα αγγλικά, γιατί μπορεί να ενδιαφέρονται κι άλλοι. Το TRS, για παράδειγμα, νομίζω ήταν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι με ρώτησαν για αυτό το σημείο. Και από αυτού θέλω να σας πω ότι η ευελιξία μας είναι πλήρης. Θα εξαρτηθεί και από το τι θα κάνετε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια πρόταση που είναι αρκετά ευέλικτη πιστεύω για να τη δούμε και υπό διαφορετικό πρίσμα. Οπότε, άμα θέλετε, ευχαριστώ Και υπήρχε και κάτι άλλο που με ρωτήσατε, σημαντικό, και μοιάζει λίγο και με αυτό που ρώτησε και η κυρία Ντάλη, το θέμα του free rider. που δεν πληρώνουν. Το ρωτήσατε και οι δύο αυτό. Οι χώροι μέλη και συνδεδεμένες συνεισφέρουν φυσικά οικονομικά στον ορίζοντα 2020, οπότε οποιαδήποτε νομική οντότητα ε, μπορεί να είναι επιλέξιμη για τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και τους πόρους που χρειαζόμαστε για την Ευρώπη και για την ε, πρωτοβουλία αυτή πρίμα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται η συνεργασία Βορρά-Νότου και πρέπει να φανεί ότι ανταποκρίνονται στους στόχους του πρίμα οι υπόλοιποι. Ακόμα και αν περιλαμβάνονται και οντότητες οι οποίες δεν ανήκουν στις χώρες οι οποίες συνεισφέρουν. και έτσι σχεδιάζεται το ετήσιο πρόγραμμα. Οι χώρες λοιπόν που δεν συμμετέχουν στο πρίμα δεν μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία. Σας το διάβασα γιατί είναι κάτι σημαντικό που θα ήθελα να καταλάβετε. Οπότε, αυτό που ρώτησε η κυρία Ντάλη για το TRL, η απάντηση είναι αυτό που σας είπα για την ευελιξία. Ήταν μια πρόταση και είμαστε ευέλικτοι να συζητήσουμε και να προσαρμόσουμε λαμβάνοντας υπόψη τα όσα είπατε. Απάντησα ήδη για το, τα διαρθρωτικά ταμεία. Νομίζω αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Όπως βλέπουμε, πολύ καλή ιδέα. Τη δέχονται οι ευρωβουλευτές και όχι μόνο οι παρόντες εδώ σήμερα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί είναι μια πολύ καλή ιδέα και για τη διαδικασία ένταξης, ε, για τη διαδικασία ολοκλήρωσης και για να βοηθήσουμε και τις γείτονες χώρες θα βελτιωθεί έτσι η κατάσταση και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά για την πρωτοβουλία σα. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, δεν ξέρω αν θα είναι φέτο ή του χρόνου, του χρόνου. καλά Χριστούγεννα τότε. Καλή, καλή Καλό χρόνο. καλή χρονιά. Να δούμε τι θα φέρουν τα... Α, α, θα έχουμε ποτό για τα Χριστούγεννα και θα καλέσουμε και τον Επίτροπο, βεβαίως. Ωραία, εντάξει, το πήρα πίσω το καλά Χριστούγεννα. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Στις 3 θα συνεχίσουμε για την διαστημική στρατηγική. Στις 3 σας ευχαριστώ πολύ.